Uh, να ξεκινήσουμε την συνεδρίαση μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Όποιος λοιπόν θέλει να καθίσει παρακαλώ. Λυπάμαι που είστε όρθιοι κάποιοι πίσω. Δυστυχώς δεν υπάρχουν θέσεις για όλους. Θα μπορούσατε ίσως να καθίσετε στα πίσω έδρανα και αν uh, σας ζητηθεί από αυτούς που δικαιούνται να καθίσουν εκεί να σηκωθείτε, να σηκωθείτε. Rose. So I would like to say on, uh, on behalf of... Εκ της Επιτροπής ε, Ρέγγι, να πω ότι χαιρόμαστε πολύ που έχουμε μαζί μας και τους συναδέλφους μας από την Επιτροπή Ήτρε για να συζητήσουμε στήματα άκρο σημαντικά, όχι μόνο για την ε, επόμενη έκδοση των πολιτικών μας για το δημοσιονομικό πλαίσιο, το πολιετές από το 2013 και μετά, αλλά όσο βουλευτές θεωρούμε ότι έχουμε και καθήκον να μην φυστούμε προσπαθειών ώστε και η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη ορίζον 2020 να συνεργαστούν, να παραγάγουν συνέργειες γιατί έτσι η Ευρώπη και θα αναπτυχθεί αλλά και θα μπορέσει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να είναι πιο ανταγωνιστική. Θα συμπροετρεύσουμε με την ε, κυρία Μάλια Σαρτόρη, την πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε, στην οποία θέλω να δώσω το λόγο για να πει και αυτή δύο λόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή Βιομηχανία ε, εκφράσει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ε, σημερινή αυτή κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, ώστε να υποδεχθούμε από κοινού τους φιλεξενούμενους για να συζητήσουμε το πιθανό μέλλον για την ε, πολιτική συνοχής. Η συζήτηση που έχει γίνει σχετικά ή και στα πλαίσια της Επιτροπής οδήγησε στο εξή συμπέρασμα. Παρότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και χρόνια, ήδη από το 2007. Είναι που, ξεκινήσαμε να συζητούμε το πώς μπορούμε να αναπνεύσουμε καλύτερα τα κονδύλια που δαπανούμε για τα ερευνητικά προγράμματα μέσω των διαφορετικών ταμείων. Και αν αυτή η συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια επιλογή, σήμερα έχει καταστεί αναγκαιότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι πλέον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απλή συζήτηση, πρέπει να ακούσουμε, να κατανοήσουμε και μετά να αποφασίσουμε πώς δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα διαθέσιμα κονδύλια από τον προπολογισμό μας και ιδίως από τα προγράμματα έρευνας και κοινοτομίας και από τα διευθυντικά ταμεία ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε ως προς το εξής. Πώς οι συνέργειες ανάμεσα σε αυτούς τους κόσμους μπορούν να δώσουν πνοή και δύναμη σε αυτή τη λέξη που την ακούμε καθημερινά ε, όλοι μας συνεχώς, για την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη όμως θα πρέπει να αποκτήσει περιεχόμενο. Θα πρέπει να μιλήσουμε για συγκεκριμένα ε, πράγματα, για να έχουμε συγκεκριμένα project και να υπάρχουν κατάλληλοι πόροι. Θεωρώ ότι η σημερινή ακρόαση Πιστεύω ότι μπορεί να δώσει συγκεκριμένε απαντήσει στο ερωτήματα. Εγώ θα είμαι μαζί σα στι τι 4. Θα ακούσω μεγάλη προσοχή όλου του ομιλητέ και ελπίζω ότι η ακρόαση αυτή θα καταστεί πραγματικά χρήσιμη. Σα ευχαριστώ. Κυρίσω λοιπόν την αξία αυτή τη ακρόαση, Μια μισή ώρα θα διαρκέσει. Έχουμε τέσσερι εξαιρετικού ομιλητέ με πολύ μεγάλη εμπειρία και ελπίζω ότι να είναι και ικανοί να μας παρουσιάσουν με τρόπο που να μας εμπνεύσει τα πράγματα. Έχουμε τον καθηγητή Γιάτση Κουγκουλίνσκι, υφυπουργό επιστημών και ανώτη της εκπαίδευσης της Πολωνίας. Έχουμε την καθηγήτρια Μπιργκίτα Βόλφ, ε, Υπουργό του Ομοσπονδίου Κουρατοδίου της Σαξονίας, Άνχαλ, τη Γίνη Αρμόδη για τα θέματα οικονομίας και έρευνα, τον κύριο Τιμ Κλέι Πόλα από το Πανεπιστήμιο Σόνση της Ουαλίας, και την κυρία Τριάννα Γκρίμη που είναι η διευθύντρια ε, του γραφείου και η επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της περιοχής της Πούλια στην Ιταλία. Θα σας παρακαλέσω να μην υπερβείτε τα 15 λεπτά, 10-12 λεπτά το πολύ ο καθένας σας, ώστε να μπορέσουμε μετά να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Πρώτον, καλώ τον κύριο καθηγητά, καθηγητή Γιάτσεκ Γκουλίνσκι να λάβει το λόγο και να μα μιλήσει για τις συνέργειες μεταξύ των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Η ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομίας ουσιαστικά ε, προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή όλων των κρατών μελών να λάβουμε υπόψη ε, τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες όλων. Πρέπει να υπάρχουν απαραίτητε δεξιότητες οι οποίες θα μεταφραστούν ε, στην ευημερία του συνόλου της ε, ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ε, ενίοτε ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά και ποικίλα εμπόδια. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδίως εν καιρό κρίσης, θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε το διανοητικό δυναμικό που είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Εάν πάρουμε έτσι λίγο απόσταση και δούμε αυτό το διανοητικό κεφάλαιο που έχουμε και στις πολιτικές έρευνας και ανάπτυξης, θα διαπιστώσουμε ότι είναι Πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη και των ε, προκλήσεων απανταχού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία θα πρέπει να διατεθούν ε, ε, τεχνολογίες εχμής και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που θα πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες οι νέοι επιστήμονες ε, να τους δοθούν περισσότερες ευκαιρίες. Βέβαια το πρόγραμμα Horizon 2020 δεν μπορεί να καλύψει όλες τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ του ορίζοντα 2020 και των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και μεταξύ του προγράμματος ορίζοντα 2020 και του έργου του προγράμματος COSME. Η επιστημονική κοινότητα άλλωστε ζητεί να υπάρξει καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων αυτών των προγραμμάτων. Αλλά ζητεί και την αύξηση του επιστημονικού δυναμικού των κρατών μελών. Άρα αύξηση και των αντίστοιχων προϋπολογισμών, 200 δις ευρώ. Εάν λοιπόν θέλουμε να υπάρξουν συνέργειες ε, μεταξύ του 7ου προγράμματος πλαισίου και άλλων προγραμμάτων και έχουν γίνει προσπάθειες και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να πω και εγώ ότι η Πολωνία έχει καταφέρει πολλά πράγματα. Έχουμε προγράμματα, έχουμε έργα που αναπτύσσουν τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών κλάδων και επιστημονικής κοινότητας. Αλλά υπάρχουν και διακρατικά προγράμματα, όπως είναι το ERANET ή το Joint Program Initiative, για να σας αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Πρέπει να εμπνευστούμε για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις. Έχουμε κάποια μέσα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα Horizon 2020, όπως το EIA δεν έχουμε υπερπηδήσει βέβαια όλα τα προβλήματα. Παραδείγματο χάρη στον τρόπο της διεξαγωγής της έρευνας. Ή δεν υπάρχει επαρκής ε, δυνατότητα, δεν υπάρχουν επαρκή σπόροι. Όλα αυτά επηρεάζουν και το ποσοστό συμμετοχής των κρατών μελών στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Το 10% των μεγαλύτερων επιστημονικών κέντρων, όπως γνωρίζετε, είναι υπεύθυνα για το 90% του συνόλου της ε, διεξαγόμενης έρευνας. Και έτσι περιφεροποιούνται άλλα κέντρα επιστημονικά. Βέβαια με κέντρα αριστείας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αν υπάρχει συνέργεια λοιπόν του ορίζοντα 2020 και με τις πολιτικές συνοχής, αυτό θα βοηθήσει να δημιουργηθούν ε, κλάστερς, ευρωπαϊκές ομάδες για την ανάπτυξη πρωτοβουλειών. Μπορούν να αναπτύσσονται με τον τρόπο αυτό υποδομές που θα υποστηρίζονται και θα χρηματοδοτούνται και από τα δύο, ε, και τους δύο αυτούς πυλώνες. Έχουμε προγράμματα όπως είναι το Marie Curie, κάποιες κοινέ ερευνητικέ δράσεις από γειτονικέ περιοχές ή περιφέρειες. Αυτά είναι πρωτοβουλίες που μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και οι συνεργασίες αυτές θα οδηγήσουν ε, και στην ε, προώθηση περαιτέρω της αριστείας αυτής ε, και την εξάπλωσή της σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, άρα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει και προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος Horizon 2020. Πρέπει να φροντίσουμε οι διατάξεις να εφαρμόζονται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Η αξιολόγηση τώρα της αριστείας των ερευνητικών προγραμμάτων και σχεδίων είναι σημαντικό γιατί θα αυξήσει την ποιότητα των ερευνητικών σχεδίων θα βοηθήσει να αξιολογηθεί καλύτερα και η εκάστοτε ομάδα, βέβαια. Η Κομισιόν έχει κάνει κάποιες προτάσεις και προβλέπει διατάξεις που όμως δεν είναι παρκείς ό,τι αφορά χάρη την εξειδίκευση ε, αυτών των κέντρων αριστείας. Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά περιφερειακών προγραμμάτων για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό, να εντοπίσουμε ποια είναι τα καλύτερα δυνατά κέντρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε διεθνή κλάστερς, να προωθήσουμε την ευφυή e e εξειδίκευση, αν μπορώ να την πω έτσι. Και όλα αυτά είναι δυνατά με τη δημιουργία συνεργειών, με την πολιτική καινοτομίας, αλλά και με την πολιτική συνοχής. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε και την διοικητική διάταξη, διάσταση, συγγνώμη. Γίνονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020. Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να εστιάσουν κυρίως ε, στην ε, διάθεση περισσότερων κονδυλίων και σίγουρα βέβαια στην εξασφάλιση της σωστής ε, δαπάνης αυτών των πόρων. Θα πρέπει επίσης τα κονδύλια συνοχή σε εθνικό επίπεδο να είναι έτσι στοχευμένα ώστε να προωθούν ε, τις διατροπτικές μεταρρυθμίσεις, να προωθούν την αριστεία και να προετοιμάζουν ε, και τις σχετικές ερευνητικές ομάδες. Μεγαλύτερη συμμετοχή επίσης σε ερευνητικά προγράμματα. Τώρα από διοικητικής πλευράς πρέπει να τακτοποιήσουμε, να διαρθρώσουμε ε, μία σειρά εκρεμή ζητήματα. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν έχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων για την ε, τον υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στα διάφορα προγράμματα. Τα Ταμεία Συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα σχετικά κονδύλια, εύκολα, πιο εύκολα διατίθεται στους δικαιούχους σε σχέση με τα κονδύλια του προγράμματος πλαισίου. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί μεταξύ πολιτικής ε, συνοχής ε, και ορίζοντα 2020. Αυτό θα αποθαρρύνει ε, την ζήτηση αυτών των κονδύλιων από τους δικαιούχους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγουμε. Πρέπει λοιπόν να εξαλείψουμε τις διαφορές αυτές και στην δημιουργία των υποδομών και αυτό που το πετύχουμε μεταξύ άλλων και με την ενθάρρυνση της συνεργασίας. Η συνεργασία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εργαλειοθήκης μας προς την αριστεία. Τα ταμεία συνοχής, τα κονδύλια συνοχής χρησιμοποιούνται ήδη για μια σειρά δράσεων που έχουν επιφέρει ήδη συνέργειες και στο πλαίσιο του ήδη φυστάμενου προγράμματος πλαισίου, αλλά και σε άλλα μέσα. Πολλές φορές ε, έχουμε εκφράσει την άποψή μας ότι θα πρέπει τα κονδύλια αυτά να διατίθενται και για τη διεθνή συνεργασία ή για συμμετοχή κάποιων ομάδων σε αμοιβαία βάση σε κάποια προγράμματα. Πρέπει να προωθηθεί η συγκρότηση διεθνών ομάδων, η βελτίωση των ε, κοινών υποδομών. σε διακρατικά προγράμματα θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή χρηματοδότηση, ένα σκέλος τουλάχιστον με κάποια καταναλογία ε, συμμετοχή. Ιδίως στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει η Μπυργκίτα Βόλφ. Α, δεν έχει έλθει ακόμη. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τότε να δώσω το λόγο στον καθηγητή Τιμ Κλέιπολ. Uh, Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είμαι ιδρυτής και γενικός διευθυντής του Τμήματος Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Σουάνση στην Ουαλία και θα σας ενημερώσω για το πώς εμείς χρησιμοποιούμε τα διευθυντικά κονδύλια και τα κονδύλια για την έρευνα για να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελος τοπικής κοινωνίας. Πρώτα απ' όλα σας μιλήσω για το ίδιο το printing. Τι είναι το printing, printing ως τύπωση. Ε, σας πάει κατευθείαν το μυαλό στα έντυπα μέσα, στις εφημερίδες και την τυπογραφία. Εγώ θα σας πω σε ότι αφορά μια πολύ μεγάλη βιομηχανία που δεν περιορίζεται στα έντυπα, αλλά ε, καλύπτει μια σειρά προϊόντων που φέρουν ε, στοιχεία τυπογραφίας, ιδιροχισμού ε, και πολλά καταναλώσιμα αγαθά αγαθά και εξαρτήματα του αυτοκινήτου σας ή ενός αεροσκάφους. Και αν αυτά σας φαίνονται περίεργα, να σας πω ότι ακόμα και τα σήματα ε, που τα φωτεινά σήματα στους δρόμους και αυτά χρησιμοποιούν αν θέλει τεχνολογία της τυπογραφίας και από την άλλη ακόμα και το μέσο της υγείας για παράδειγμα για την παραγωγή της σωμάτων. Άρα λοιπόν για την ε, έρευνα χρησιμοποιείται πέρα από πολύ πολύ τεογραφία. Αυτό το printing που λέω λοιπόν, είναι λοιπόν μια βιομηχανία τεράστια που μπορεί να δώσει πάρα πολλά αποτελέσματα. Κατανοείται λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια δραστηριότητα που καλύπτει μια σειρά παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ακόμα και το ε, τύπο νομίσματος, ε, διαβατηρίων, ε, λοιπόν εγγράφων. Αλλά αυτό αφορά ακόμα και τα άκρα, τα ανθρώπινα άκρα. Πώς γίνεται αυτό, μα για την αντικατάσταση σε περίπτωση ατυχήματος. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια μηχανία που κυρίως αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσει όσο να σα φαίνεται περίεργο. Σε ό,τι αφορά την συσκευασία και τα έντυπα, μιλάμε για 123.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 18.500 ε, ανθρώπους ε, στην τοπική βιομηχανία. Κυρίως πρόκειται για μια βιομηχανία που πιο πολύ έχει τεχνικά χαρακτηριστικά. Πριν λαμβάνουμε κονδύλια από τα διευθυντικά ταμεία ή εργαζόμασταν στενά με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και θα έλεγα ότι το περίεργο στοιχείο είναι ότι έχουμε πιο μεγάλο αντίκτυπο ε, εκτός της Ουαλίας και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ε, είχαμε μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ΙΠΑ ε, και σε άλλα μέρη του κόσμου και όχι σε ένα χωριό ε, κοντά στο πανεπιστήμιό μας, στην Ουαλία. Χρησιμοποιούμε πάντως τις δυνατότητες μας δύνατα για να διαρθρώσουμε, αν θέλετε, την έρευνά μας παράλληλα με τις τοπικές ανάγκες διορίσαμε έναν Ευρωπαίο αξιωματικό σύνδεσμο για να μας ενημερώνει καλύτερα τι είναι τα ταμεία. Εγώ δεν είχα ιδέα τι είναι τα ταμεία. Αυτή η αξιωματικό σύνδεσμο που με ρώτησε, μα γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου, γενικότερα των ταμείων, για να στηρίξουμε αυτές τις δραστηριότητες και να κάνουμε τη μεταφορά της γνώσης. Να χρησιμοποιήσουμε το κοινωνικό ταμείο για την εκπαίδευση για την κατάρτιση, διότι αν κανείς κινείται από μια βιοτεχνική δραστηριότητα σε μια βιομηχανία υψηλής ε, τεχνολογίας, χρειάζεται τέτοιου είδους κονδύλια. Επίσης χρησιμοποιούμε το κοινωνικό ταμείο για ε, μεταπτυχιακές σπουδές. Έπειτα χρησιμοποιούμε το τύπο ένα ακρονίμιο για κάθε εφαρμογή. Το τύπο λοιπόν είναι μια εφαρμογή για την έρευνα εχμής για όλο τον κόσμο που γίνεται προ όφελο μουσεών επιχειρήσεων και κέρδισε και ένα βραβείο το 2009 για αυτή την επιχειρηματικότητα. δραστηριότητα. Θεωρούμε ότι για να υπάρχει επιτυχία πρέπει να έχουμε μια ε, στρατηγική περιφέρεια που επιλέξαμε και να γνωρίσουμε τι απαιτεί η βιομηχανία. Αυτή τη γνώση την αποκτήσαμε μέσα στα χρόνια από τι διάφορε εθνικέ δραστηριότητε και το σύνδεσμό μα με τι πολυεθνικέ επιχειρήσει. Επίση, χρειαζόμαστε ακαδημαϊκού που του ενδιαφέρει να γράφουν άρθρα στι εφημερίδες αλλά και να αναπτύσσουν project παράλληλα με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Είχαμε πολύ σημαντικό κύκλο εργασιών αυξάνοντας το κύκλο εργασιών κατά 5 εκατομμύρια ε, ευρώ σε ό,τι αφορά τις εταιρείε με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Πώς θα συνδέονται με το θέμα που συζητούμε, χρησιμοποιούμε τη δεκαταμία για να δημιουργήσουμε καλύτερη υποδόμηση δυναμικού ε, είμαστε πιο σειρή θέση για να ε, αποσπάσουμε κονδύλια από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας. Επίσης ε, δίνουμε καταστάσεις, ε, μάλλον πρόσβαση σε καταστάσεις για όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Επίσης είμαστε ένας κόμπος, ένας κέντρος για, τα, για την έρευνα στα ηλεκτρονικά και επίσης ανοίγουμε νέους δρόμους για να μπορέσουμε να κάνουμε ε, κοινή έρευνα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, έρευνα για τη ταχύτερο ε, φως, για παράδειγμα την εταιρεία Philips, κάνουμε σχετική έρευνα σε όλη την Ευρώπη και έχουμε και άμεση που είναι ένα καινοτόμο πρόσβητο που ε, ηγούνται σε αυτό. Ε, επιχειρήσεις για την ταχύτερη πούλωση τραυμάτων. Τώρα, προκλήσεις. Εγώ θα εστιάσω στα θέματα υπογραφής γιατί αυτή είναι η δική μου δουλειά. Τι ευκαιρίες μπορούμε να δούμε. Προηγμένη μεταποίηση με τυπογραφία, έξυπνη συσκευασία και α, πρόοδο και στον τομέα της υγείας, στα ανθρώπινα άκρα, όπως είπα, που μπορούν να μας εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια ευρώ ε, ετησίως. Και μιλάμε για ένα άνοιγμα σε πολύ μεγάλες αγορές. Κάτι άλλο που γνωρίζουμε είναι ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, αλλά μέσα στην Ευρώπη υπάρχουν και άλλα ερευνητικά κέντρα εχμής με τα οποία θέλουμε συνεργασία. Αν θέλουμε μια στρατηγική για την Ευρώπη, χρειαζόμαστε να είμαστε σίγουροι ότι ο Horizon 2020 διασφαλίζει ε, ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της έρευνας και της επιτρέπει επίσης ε, να ε, θέλει σε πιο είναι συνεργασία τους ερευνητές. Χρειάζονται λοιπόν ερευνητικά κονδύλια σε αυτό το σκοπό. Ό,τι αναπτύξαμε ε, στο παρελθόν, το εκμεταλλεύτηκαν πιο πολύ η και το Σουόνσι. Και δεν καταφέραμε να ε, λειτουργήσει αυτό προς όφελος της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χρόνια τώρα ξέρουμε ότι είναι πρωταθλητή στο Σουόνσι για την καλή χρήση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τώρα καταλαβαίνω καλύτερα. Ε, μάλλον βλέπω ότι και η κυρία Μπριγκίτα Βόλφ είναι μαζί μας. Αν θέλετε να σας δώσω το λόγο να κάνετε την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που άργησα. Νομίζω ότι στα γερμανικά θέλετε να κάνετε την παρουσίαση. Είμαι από την ε, Σαξονία, ένα από τα νέα κρατήδια της ε, Γερμανίας και είμαστε, αν θέλετε, μια περιφέρεια υπόδειγμα κατά κάποιο τρόπο για αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε εδώ σήμερα. Και αυτή είναι μια περιφέρεια υπόδειγμα. Η Ανατολική Γερμανία εδώ και 20 χρόνια σε ό,τι αφορά την επιστήμη και την έρευνα. Είμαστε λοιπόν υποδειγματικοί και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο της Δυτικής Γερμανίας. Φυσικά η το σημείο εκκίνησης μετά από 40 χρόνια σοσιαλισμού δεν ήταν συγκρίσιμο με την υπόλοιπη Γερμανία. Άρα ως εκ τούτου εποφεληθήκαμε και ε, από την ε, Δική Γερμανία και από την Ευρώπη. Ήμασταν περιφέρεια ε, στόχου 1 και προσπαθήσαμε και με την κατάλληλη ε, χρήση των ευρωπαϊκών μέσων να αναπτύξουμε την έρευνα και την επιστήμη, την οποία και συμπληρώσαμε μετά με τα δικά μας ε, κρατικά μέσα, για αυτό που ονομάσαμε Staircase to Excellence, σκάλα προς την αριστεία. Αυτό προσπαθήσαμε να διοργανώσουμε. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για μας, αλλά και για άλλα κρατήτια της Ανατολικής Γερμανίας. Παρόμοια κινηθήκαν και αυτά. Δεν είμαστε ακόμη στην κορυφή της ε, κλίμακας, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε πολλά τα τελευταία 20 χρόνια. Πολλά ε, ευρωπαϊκά διερφωτικά κονδύλια λάβαμε και αυτό μας βρίσκει ευγνώμονες την πρώτη περίοδο 1,93 δισεκατομμύρια ευρώ, την δεύτερη περίοδο πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και Υποστηρίξαμε 1.300 σχεδόν ε, project, έργα. Τα πιο πολλά εξ αυτών εστιάζονται στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Στα πανεπιστήμια μας έχουμε περίπου 32.000 ε, Έχουμε ταπανίσει 31.000 ε, εκατομμύρια Τώρα να σας πω τι εννοώ με το Staircase to Excellence. Ε, ένα πρώτο παράδειγμα. Είχαμε μία παράδοση σε ό,τι αφορά την, ε, τις νευροεπιστήμες. Ε, Μην με ρωτήσετε τι ακριβώς σήμαινε αυτό στην Ανατολική Γερμανία, αλλά ήταν καλή, καλό το σημείο εκκίνησης. Το 2001 λοιπόν η κυβέρνηση του κρατηδίου αποφάσισε με μέτρα με μέσα του κρατηδίου αλλά και με ευρωπαϊκά μέσα να δημιουργήσει το πρώτο σπιθρογράφημα και την πρώτη σχετική συσκευή. Και από το 2002 και μετά λοιπόν, ε, χάρη στα ευρωπαϊκά αυτά μέσα, καταφέραμε να προάγουμε αυτά τα μέσα, αυτές τις συσκευές. Βλέπετε λοιπόν ότι χρησιμοποιήθηκαν και οι πανεπιστημιακές ε, δυνάμεις και μόνο με την ειδική αυτή συσκευή καταλαφέραμε να δώσουμε τη δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα και αυτό αποτέλεσε τη βάση για το Εθνικό μας Ίδρυμα Έρευνας και έτσι όλο και πιο πολύ καταφέραμε να ε, καταρτήσουμε και τους νέους επιστήμονες. Και αυτό εννοούμε με την κλίμακα προς την αρεστία. Το 2006 αποφασίστηκε να δημιουργηθεί το κέντρο για την ε, ε, συμπεριφορική ευρωεπιστήμη. Δεν είναι μόνο οι ψυχολόγοι και οι ιατροί που εργάζονται σε αυτές τις ε, εγκαταστάσεις. Εργάζονται κοινωνικοί επιστήμονες ειδικοί σε κοινωνικά θέματα ειδική σε θέματα IT και έτσι μέσω της ορατότητας και της κρίσιμης μάζας που έχει συγκεντρωθεί καταφέραμε να καταρτήσουμε τον τομέα αυτό ένα επιτυχημένο τομέα. Ένα επόμενο σημαντικό βήμα έγινε το 2012. Τώρα λοιπόν δεν προέκυψαν φυσικά όλα αυτά σήμερα, αναπτύχθηκαν σταδιακά. Έχουμε στο Μάκτεμπουργκ το Ινστιτούτο Λάιπνιτς για την νευροβιολογία για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Και βλέπετε πώς από ε, ένα μικρό θύλακα καλών επιστημόνων με τη σωστή δομή και διάρθρωση μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο κέντρο. Και εντωμεταξύ οι ερευνητές της ομάδας αυτής έχουν ενταχθεί στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και σε πολλά προγράμματα συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες, με τη Siemens, αλλά και με πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεργάζονται με όλες αυτές και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νευροεπιστήμες και με την τεχνολογία την ιατρική υπάρχει ε, μια ελπίδα, γιατί ξέρετε υπάρχει γενικώ ένα κενό στα θέματα αυτά στην υπόλοιπη Γερμανία στην υπόλοιπη Δυτική Γερμανία. Άρα λοιπόν αυτό αποτελεί ε, μια, ένα δυνατό μας ε, σημείο. Κάναμε και διάφορες ε, έρευνες σε άλλα κρατήδια και βλέπουμε ότι έχουμε και πάρα πολλά ιδρύματα Max Planck, ιδρύματα Leibniz, ακριβώς για να πλαισιώσουν αυτή την ανάπτυξη και αυτό φαίνεται ότι ε, έχει αρχίσει και να γνωρίζετε το κύρος μας σε όλη τη Γερμανία. Να σας δείξω και μερικά άλλα παραδείγματα και αυτού του έργου αλλά και άλλων έργων. Βλέπετε για παράδειγμα τον πρώτο πινθυρογράφο το νέο Ινστιτούτο, το νέο Ίδρυμα που δημιουργήθηκε φέτος και γι' αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά διαφορετικά ταμεία, αλλά έχουν απασχοληθεί και πάρα πολλοί ευφυείς ε, άνθρωποι, τους οποίους μπορέσαμε να προσελκύσουμε ακριβώς επειδή είχαμε το κέντρο αυτό. Το επόμενο βήμα θα είναι να δημιουργηθεί το τσίκλοτρον. συνεργαζόμαστε στενά με τη Siemens προς την κατεύθυνση αυτή. Και εδώ έχουν δαπανηθεί πολλά κονδύλια και κονδύλια των ε, διευθυντικών ταμείων για την ανάπτυξη ε, προϊόντων που θα μπορούν να διατεθούν στην αγορά σε ό,τι αφορά το κυκλοτρόνιο αυτό. Ένα άλλο θέμα το οποίο προηθούμε, το Magdeburg, ήταν μετρόπολη για ε, μεγάλα μηχανήματα. Προσπαθούμε λοιπόν από την παράδοση αυτή να ωφεληθούμε και για την ε, κατασκευή αυτοκινήτων. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ε, δαπανηθεί ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που θέλουμε, αλλά έχει γίνει πολλή δουλειά. Επίσης κάτι άλλο, σε ό,τι αφορά το engineering και το virtual development, ένα κέντρο για την ε, εικονική ανάπτυξη και κατάρτιση, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Και εδώ έχουν δαπανηθεί ευρωπαϊκά κονδύλια στον τομέα της βιοτεχνολογίας, το νότο του κρατηδίου μας έχουμε σημειώσει κάποια επιτυχία. Ε, παραδοσιακά έχουμε ε, ιδιαίτερα αναπτυγμένο χημικό κλάδο και έχουμε και φυσικούς πόρους που υποστηρίζουν ε, την ανάπτυξη αυτή και αυτά ε, πάντα φυσικά και με ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και με συγχρηματοδότηση από το κρατήδιο και από το κράτος της Γερμανίας. Ε, να κάνω λοιπόν να εξαγάγω κάποια συμπεράσματα. Η εμπειρία μας είναι ότι έχει λειτουργήσει, ότι μπορούμε μέσω της ε, αξιοποίησης, της συμπληρωματικής αξιοποίησης των στρατικών ταμείων να δημιουργήσουμε υποδομές. υποδομές φυσικά, τα όμορφα κτίρια χωρίς τα ανάλογα μυαλά δεν αξίζουν τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά όπου μαζεύεται η κρίσιμη μάζα τελικά μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Και εδώ σε αυτό το σημείο μπορεί να είναι καθοριστική η σύμβολη των διαρθωτικών ταμείων. Γιατί κάποια πράγματα πολύ απλά δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε μόνοι μας. Άρα έχουμε πάρα πολύ καλά παραδείγματα και πολύ καλές εμπειρίες ε, μέσω της συμπληρωματικής αυτής της χρηματοδότησης. Αναέφερα ήδη ότι η υποδομή καθιστά πιο εύκολο να προσελκυθούν εξαίρετοι επιστήμονες σε, μια, ε, σε ένα περιβάλλον το οποίο κατά τα άλλα μπορεί να μην εμπνέει ιδιαίτερα κορυφαίοι επιστήμονες δηλαδή οι οποίοι έχουν εργαστεί σε διεθνώς καταξιωμένα ε, ιδρύματα Max Planck, για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία, στην ΗΠΑ. Ε, πολλοί επιστήμονες επέστρεψαν στην Ανατολική Γερμανία και συνέχισαν την έρευνα του. Σε πολλές περιπτώσεις έφεραν μαζί και την ομάδα τους. Αυτό ακριβώς θέλαμε να πετύχουμε. Θα προσέξατε ότι στην παρουσίασή μου συχνά αναφέρονται ερευνητικά κέντρα όπως το Max Planck, το Fraunhofer, το Leibniz, το Heinholz στη Γερμανία. Αυτά είναι τα μεγάλα έξω πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα και αυτά τα κέντρα στην ανάπτυξη της Ανατολικής Γερμανίας έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό με οδηγεί στη σκέψη του teaming και twinning που επίσης έχει προταθεί. Έχουμε πάρα πολλές καλές, πολύ καλές εμπειρίες σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θηγατρικών, αν θέλετε, ιδρυμάτων όπως αυτά του Max Planck και κάποια από αυτά έχουν δημιουργηθεί ως spin-offs, ως ε, θηγατρικές ε, τέτοιων ε, δυτικών ιδρυμάτων στο νότο του κρατηδίου μας και αυτό μας βοήθησε γιατί ξέραμε ότι τεχνικά ήμασταν σε σωστό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι η ιδέα του teaming, and twinning, δηλαδή η δημιουργία ομάδων και η αδελφοποίηση, αν θέλετε, των ιδρυμάτων, είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Εμείς στη ε, Σαξονία Ανχάλτ ε, εποφεληθήκαμε ασφαλώς και θα θέλαμε και θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα ασφαλώς αν στο μέλλον ε, μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να βρούμε άλλες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και τώρα να δώσω το λόγο στον, ε, στην κυρία Αντριάννα Αγκρίμη από την περιφέρεια της Πούλια. Έχετε το λόγο. Ε, ε, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει στην περιφέρεια της Απουλίας. Και η μαρτυρία που έχουμε μας επιτρέπει να προτείνουμε ένα συγκεκριμένο εργαλείο για να πετύχουμε το στόχο της συνεργίας ανάμεσα στον ορίζοντα 2020 και τα διεθνωτικά ταμεία. Αυτό το εργαλείο λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, είναι το Smart Specialization, η έξυπνη εξειδίκευση, η ικανότητα, αν θέλετε, των περιφερειών να οικοδομήσουν, υλοποιήσουν και να παρακολουθούν μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης ε, σε τοπικό επίπεδο, ώστε να λαμβάνει υπόψη διαρθρωμένα τις δυνατότητες που δίνει και ορίζοντας 2020 και τα Η περιφέρεια της Απουλίας χρησιμοποιεί τα κατά μία, κατά κύριο λόγο για την επίτευξη αναπτυξιακών ε, στόχων ε, στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και θα συνοψίσω ε, εντάχει αυτούς τους στόχους γιατί δεν είναι νομίζω ότι εδώ το κατάλληλο βήμα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αναφέρω όμως ένα παράδειγμα πιο συγκεκριμένα για να σας δώσω ένα παράδειγμα των πιθανών κατά τη γνώμη μας συνεργειών ανάμεσα στα αγροτικά ταμεία και τον Ιούς το 2020. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ότι απαιτείται μία στρατηγική για την έξυπνη χρήση των κονδυλίων, των ταμείων. Αν δεν υπάρχει μια τέτοια έξυπνη στρατηγική για ολοκληρωμένη χρήση των ταμείων, τελικά δεν θα έχουμε αποτελεσματικότητα. Αυτή είναι η προσέγγιση που κρίναμε σκόπιμο να ακολουθήσουμε. Ώστε κάθε γραμμή παρέμβασης, όπως εδώ βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια, να συνδέεται άρρηκτα με τις υπόλοιπες, ανεξάρτητα από τη φύση των χρησιμοποιούμενων ταμείων και από την κλίμακα παρέμβαση. Είναι μια κλίμακα που ξεκινά από το περιφερειακό επίπεδο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το περιφερειακό ε, επίπεδο και φτάνει το ευρωπαϊκό. Στη δική μας περιφέρεια, στην περιφέρεια της Απουλίας, η λέξη κλειδί είναι η κρίσιμη μάζα, η δημιουργία δικτύων, η δημιουργία συνδέσμων και η δικτύωση ανάμεσα στους φορείς. Και ιδιαίτερα η εστίαση πέφτει αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη κλάστερς που υπόσχονται πολλά στον τομέα του εξυγχρονισμού ή τον απεριορισμό των θέσεων των παραδοσιακών κλάστερ. Πιο πολύ λοιπόν αυτό, όπως η τον απεριορισμο των νοθέσεων των παραδοσιακων κλαστερ πιο κλάστερ σε υψηλή ένταση γνώσης. Κάποια από τα κλάστερ που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια είναι αυτά που κατά τη γνώμη μας, για τα οποία μάλλον κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να υπάρξει ε, μία κατάλληλη στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση. Αυτή η στρατηγική συνοδεύεται από την ικανότητα της ίδιας περιφέρειας να σταθεί ευρωπαϊκά σε σχέση με άλλους ευρωπαίους εταίρους, με άλλες περιφέρειες και θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη στρατηγική αυτή για να μπορέσουμε να συνοδεύσουμε τους φορείς αυτού του περιφερειακού ε, έξυπνου, αν θέλετε, συστήματος για να ε, έχουμε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο έρευνα και καινοτομία στα πλαίσια του ΡΙΖΟ 2020. Υπ' αυτή την έννοια προσπαθούμε να δημιουργήσουμε να αναπτύξουμε μάλλον τις προτάσεις ε, δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθώντας για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε την European Innovation Partnership καθώς είναι μια πρωτοβουλία που λαμβάνει υπόψη το περιφερειακό επίπεδο Ταυτόχρονα όμως ε, και τους παραγωγικούς ε, και ερευνητικούς ε, περιφερειακούς φορείς. Το σημείο, το θέμα για το οποίο σήμερα καλούμαστε να εκφράσουμε τις θέψεις μας, που είναι δηλαδή οι συνέργειες ανάμεσα στον ορίζοντα 2020 και τα ταμεία, κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα που έχει διάφορες αποχρώσεις και αλογεύουν διάφοροι κίνδυνοι για να υπάρξουν διαφωνίες και συγκρούσεις. Από τη μία ορίζον 2020 θα επιβραβεύσει την αριστεία. Από την άλλη, τα διευθυντικά ταμεία θα πρέπει και επιθυμούν να εγγυηθούν, αν θέλετε, την ανάκτηξη ενός κοινωνικο-οικονομικού χάσματος ε, των περιφερειών η αυτή την έννοια είμαι της γνώμης ότι ο στόχος που θα πρέπει να επιτύχουμε εντοπίζοντας και ορίζοντας τις στρατηγικές είναι ο στόχος αριστείας να πρέπει να επιτευχθεί. Είναι κάτι αναγκαίο για το σύστημα της Ευρώπης. Δηλαδή θα πρέπει η Ευρώπη να στοχεύει στην αριστεία με στόχο τη διεθνή αντιγωνιστικότητα. Από την άλλη είναι εξίσου σημαντικό να δημιουργήσουμε και ε, ενάρετα, αν θέλετε, κυκλώματα, δίκτυα που να στηρίξουν αυτές τις αριστείες στην πράξη. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, αυτές οι συνεργές θα πρέπει να ε, βασιστούν στις στρατηγικές. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε, να χαράξουμε ειδικέ ε, στρατηγικές έξυπνες εξειδίκευσης των περιφερειών. Και σε αυτή την ευκαιρία ε, μας καλούν και έντονα να κινηθούμε τα ιδρυτικά ταμεία, ώστε να έχουμε εξειδικεύσεις από τη μία και συμπληρωματικότητες μεταξύ των περιφερειών από την άλλη. Μια συμπληρωματικότητα απαραίτητη, ώστε να, να δημιουργηθεί απαραίτητη κρίσιμη μάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επιτύχουμε την αριστεία. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώ ότι στόχοι και οι συνέργειες σε υπηρεσιακό επίπεδο κινούνται σε δεύτερο επίπεδο. Αντίθετα, είναι βασικό και απαραίτητο πρώτο βήμα να ασπαστούμε και να συμφωνήσουμε σε αυτή τη γενική αρχή. Συμπληρωματικότητα των ερευνητικών δράσεων. Αυτό απαιτεί μια ειδική προσοχή που πρέπει να δοθεί όχι μόνο στα νέα εργαλεία και σε νέες φόρμουλες συνεργασίας, αλλά θα είναι μια συνεργασία που θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ε, θεσμική ικανότητα των ε, πολιτικών που χαράσουν πολιτική να μεταφέρουν αυτά σε περιφερειακό επίπεδο. Μόνο έτσι τα εργαλεία γνώσης και της εργασίας ε, θα μπορέσουν να, να περαστούν να περάσουν συγγνώμη σε περιφερειακούς φορείς και να δώσουν αποτελέσματα. Υπ' αυτή την έννοια, θέλω να πω ότι εμείς αμέσως ασπαστήκαμε μία πρωτοβουλία της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΡΕΚΙΟ, την Smart Specialization Platform, που διαχειρίζεται το ε, Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της ε, Σεβίλης, γιατί μας δίνει μια σαφή και αυτή η ε, εικόνα της κατάρτισης μέσω της μάθησης, της κατάρτισης μέσω της Αξιολόγηση ομοτήμων. Είναι μια διαδικασία που προβλέπει πολλά βήματα και άρα δημιουργεί τις κατάλληλες συγκροματικότητες που κατά τη γνώμη μου θα επιτρέψουν στις περιφέρειες να πετύχουν τους στόχους του ορίστου 2020 ενισχυόμενες από τα διαφορετικά κονδύλια. Είναι σαφές ότι για τον καθορισμό και τη χάραξη αυτών των στρατηγικών ευκταίο θα ήταν ορίζοντας 2020 να επιτρέπει στις περιφέρειες να κοιτάξουν και ε, έξω από τα πλαίσια καταστήνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβουν υπόψη με μεγαλύτερη ουσία τη διεθνή διάσταση. Σε ό,τι αφορά και πάλι τις στρατηγικές, ακόμη πιο χρήσιμο θα ήταν, θα έλεγα, να υπάρχει δυνατότητα να συνεχίζεται η παρακολούθηση και η βελτίωση αυτών των στρατηγικών βάσει ενός σχήματος που δεν προβλέπεται ε, στον ορίζοντα 2020 που είναι οι περιφέρειες για τη γνώση. Ήταν ένα εργαλείο αυτό πολύ αποτελεσματικό κατά τη γνώμη μας και ελπίζουμε να μας επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο και στον ορίζοντα 2020 παραλαμβάνω ότι είναι ένα εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι περιφέρειες για να συνεχίσουν να παρακολουθούν και να βελτιώνουν στρατηγικές τους. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και εφαρμογή, υλοποίηση. Υλοποίηση ε, υπό το ευρωπαϊκό πρίσμα. Χρειάζεται λοιπόν από κοινού να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία καθαρά στρατηγικού χαρακτήρα όπως είναι το Eranet, όπως και χρήση από την άλλη διευθυντικών ταμείων για να τροφοδοτηθούν αυτά τα προγράμματα αυτό, κατά τη γνώμη μας, θα μας έδινε ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ώστε να έχουμε ε, αν θέλετε, προγράμματα και στρατηγικές ε, που να στοχεύουν ε, στην έρευνα και την κοινοτομία χρησιμοποιώντας την έξυπνη εξειδικεύση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δώσουμε, να λάβουμε υπόψη μάλλον και τη μεσογειακή διάσταση και την διεθνή επιτα διάσταση για αυτά τα θεματολόγια που θα σχηματιστούν. Από εκεί πέρα, συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων. Επί της ουσίας, κατά τη γνώμη μου, αυτό έγκυται στην ικανότητα οι παρεμβάσεις να είναι ακόλουθες και ολοκληρωμένες μεταξύ τους. Θα δώσω ένα παράδειγμα σε περιφερειακό επίπεδο που αναλογικός πώς ε, ε, ταιριάζει με την εμπειρία της αξονίας είναι οι μεγάλες ε, υποδομές σε μεγάλες περιφερειές. Να πω 40 εκατομμύρια ευρώ θα επενδύσαμε μάλλον στην Απουλία για την δημιουργία τέτοιων ε, δικτύων, ε, το δημόσιο τομέα για την έρευνα και με βάση αυτές τις υποδομές σκεφτήκαμε ότι είναι καλό, μάλλον σε αυτές τις υποδομές, να σκεφτήκαμε να κάνουμε παρεμβάσεις από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο ώστε να δούμε τον ε, τοπικό αντίκτυπο, δηλαδή τον αντίκτυπο στους γραμμαστές επιχειρήσεις, ώστε μαζί με τις γραμμαστές επιχειρήσεις της Απουλίας να κατακτήσουμε συγκεκριμένα ε, project. Αυτό το μείγμα στρατηγικής ε, διαχείρισης, αν θέλετε, μπορεί να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις δραστηριότητες ΕΣΦΡΙ και ε, στις δραστηριότητες του ΡΙΖΑ 2020. Χρειάζεται όμως να έχουμε πλήρη γνώση και κατανόηση του γεγονότος ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το βέλιο στο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο κεφάλαιο. Δηλαδή να έχουμε ε, υπόψη μας μηχανισμούς ε, που θα επιτρέψουν να υλοποιήσουμε αυτές τις ε, δραστηριότητες χρησιμοποιώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο με τον καλύτερο τρόπο. Από εκεί πέρα υπάρχουν ε, και άλλα πράγματα όπως είναι οι κανόνες, η εναρμόνιση των οικονομικών κανόνων είναι κάτι χρήσιμο. Θεωρώ ότι ίσως και να θεώρησε των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση της αριθμής κοινοτομίας ήταν κάτι χρήσιμο, ώστε να δούμε γενικότερα το θέμα της καινοτομία στα πλαίσια του Open Innovation και της δημιουργικότητας. Μια σειρά εργαλείων που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται στις περιφέρειες, όπως είναι το Living Lab, ε, ώστε να καθοδηγηθούν οι χρήστες περισσότερο, όπως και οι δημόσιες προμήθειες και οι υπηρεσίες για την καινοτομία, είναι όλα εργαλεία που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να έχουν περισσότερο χώρο στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, δύο ακόμη πτυχές ε, της ε, διαλειτουργικότητας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα δύο προγράμματα. Από τη μία θα πρέπει να επιβραβεύει ο ορίζοντας 2020 πρωτοβουλίες εκείνες που συνδέονται άρρηκτα με τις ε, δραστηριότητες έξυπνης εξειδίκευσης και καταδεικνύουν τη συμπληρωματικότητα από την άλλη για τις περιφέρειες ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρξει μια ιστροή πληροφοριών σχετικά με τη συμβολή των περιφερειακών φορέων στα ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκής κλίμακας ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να υλοποιήσουμε και να παρακολουθούμε και να βελτιώσουμε τις μα στρατηγικέ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, uh, Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Αγκρίμη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να παρακαλέσω όλου του συναδέλφου που θέλουν να λάβουν το λόγο να σηκώσουν το χέρι του τάχιστα για να υπολογίσω αν θα έχετε το καθένα 10 δευτερόλεπτα ή ένα λεπτό. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε παντός επιστητού, αλλά να υποφεληθούμε της εμπειρίας ε, των ε, επαγγελματιών που είναι εδώ. Οπότε καλύτερα θα ήταν να τους ζητήσουμε να μας ε, επιβεβαιώσουν πράγματα, να τους κάνουμε ερωτήσεις και να δούμε τι πρακτικές ανάγκες υπάρχουν ώστε να μπορεί να υπάρχει συνεργασία αυτών των πολιτικών. Είναι μια χρονική στιγμή, άλλωστε, όπου κατ' ουσίαν να συντάσσουμε τροπολογίες ε, για τις προτάσεις που έχει διατυπώσει η Κομισιόν σε σχέση με τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές. Άρα είναι η ώρα που πρέπει και εμείς να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που λείπει ή τι χρειάζεται ίσως να αλλάξει στην πράξη με βάση τα όσα ακούσαμε. Ο κύριος Γκλάντ από την Επιτροπή Τρίνο πρόσφατα το λόγο. Σας ευχαριστώ. Μία συγκεκριμένη ερώτηση έχω να κάνω. Για να απαντήσω και στην κυρία Βόλφ. Εγώ είμαι από το κρατήριο του Μπράντεμπουργκ, όπου δημιουργήθηκαν αυτά τα κλάστερ ιδρυμάτων. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα για τα ε, μέσα ε, διευθυντικών ταμείων και πώς αξιοποιήθηκαν. Αυτό που θέλαμε εμείς είναι το εξή ότι καταρχάς θέλουμε να προωθήσουμε την αριστεία στην Ευρώπη, την αριστεία στην κοινοτομία και στην έρευνα, αλλά από την άλλη και περιφέρειες που δεν είναι σε θέση να προσελκύσουν ανθρώπινο δυναμικό, να μπορούν και αυτές να ασκήσουν αυτή την άριστη έρευνα. Όταν λοιπόν κάποιος ε, ξεκινάει ε, μια τέτοια, ένα τέτοιο ίδρυμα, θα πρέπει να εγγυόμαστε ότι μπορεί να συνεχίσει, ε, για παράδειγμα, με τα προγράμματα Marie Curie, να συνεχίσει την δραστηριότητα αυτή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ε, ανταγωνισμός, δεν γίνεται να υπάρχει παντού. Να υπάρχουν παντού τέτοια ερευνητικά κέντρα. Δεν επαρκούν τα μέσα μας για την ε, σκοπό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φανδίστεροι από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ε, ευκαιρία αυτή για την ακρόαση. Αυτή βρισκόμαστε σε μια θέση που δεν είναι ανταγωνιστική μεταξύ των Επιτροπών. Προωθεί την ε, οικονομία της γνώσης και την επένδυση στην ανάπτυξη. Τρεις ερωτήσεις έχω να κάνω προς τους τέσσερις εμπειρογνώμονες. Ποια ήταν τα βασικά εμπόδια, γιατί όλοι αποδείξατε ότι τα καταφέρατε, δεν ναι. Μας εμποδίζει η νομοθεσία, ειδικά. Όχι, είναι πιο πολύ το όραμα της κάθε περιφέρειας που θέλει να επενδύσει. Κατά δεύτερον, είδατε τις νέες προτάσεις. Μιλήσατε για εξειδίκευση της αγοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σαφές και έχετε δίκιο ότι δεν μπορούμε να υπάρχουμε διπλές, ε, διπλές τέτοιες έρευνες. Θα πρέπει να συνδυάζεται πολιτική bottom-up, από κάτω προς τα πάνω στην περιφερειακή πολιτική, αλλά και από πάνω προς τα κάτω. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Και τρίτον, σήμερα το πρωί παρουσιάσαμε το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, όπου ορίζονται συγκεκριμένα τα μέσα και πώς θα μεταφραστεί η νομοθεσία για τις συνέργειες μεταξύ των δύο ταμείων. Επίσης εισάγαμε μία υποχρέωση σε όλη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά το Ταμείο ε, Διευθυντικών Ταμείων όπου θα πρέπει το 1-10% να δαπανάται εκτός της χώρας, να μην ε, κοιτούν δηλαδή μόνο το ιστορικό τους οι περιφέρειες, αλλά και το εξωτερικό. Αυτό ε, είναι μια πρόσθετη πρόταση την οποία και κάναμε πριν από κάποιες εβδομάδες. Θέλετε να σχολιάσετε παρακαλώ, μάλιστα, να ακούσουμε και τον Κρίστιαν Έλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο θέματα. Να τονίσω ότι σε όλες τις συζητήσεις, σε ό,τι αφορά αυτή την κλίμακα προς την αριστεία, ε, αυτό προϋποθέτει μια πολιτική συμφωνία όλων των πολιτικών δυνάμεων. Θυμάμαι ότι όταν είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο, ε, τότε πρόεδρο του Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου κύριο Μπούζεκ, για να συνάψουμε συμφωνίες και συμβιβασμούς για τον ορίζοντα 2020 και τότε είχε ζητηθεί να υπάρχει να γίνει διαπραγμάτευση με ποσόστοση για τις νέες ε, χώρες μέλη. Και αυτό μας είχε οδηγήσει στην εξή δύσκολη θέση. Αναγκαστήκαμε τότε να μείνουμε στην αρχή της αριστείας και είχαμε πει τότε ότι θέλουμε το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο θα διέπεται από τις παραμέτρους αριστείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιήσει το δυναμικό του. Και να δώσω ένα παράδειγμα και ίσως να ρωτήσω πώς θα πρέπει να διατυπωθεί συγκεκριμένα. Με αυτό το Stairway to Excellence και ε, με αυτή την συνέργεια μεταξύ των δύο ταμείων, πώς μπορούμε να κινηθούμε. Τα πιο, οι πιο μεγάλες επιτυχίες προέρχονται από τα κλάστερ έρευνας, επιστήμης, που ορισμού δεν χαρακτηρίζονται μόνο από αριστεία, αλλά και από μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, πυκνότητα επιστημόνων και ικανότητα συμμετοχής ε, στο παγκόσμιο προσκήνιο και ανταγωνιστικότητα. Αυτό που πάντα λείπει, ιδιαίτερα στις ε, νέες χώρες μέλη, η έρευνα και η αριστεία περιορίζεται από την διαχείριση της αριστείας και αυτό σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε την αιτία ε, για την οποία δεν συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά ταμεία. Νομίζω ότι μπορεί να συνδεθούν λοιπόν τα διαφορετικά ταμεία με τον Ρίζοντο 2020. Πρόκειται για ομίλους οι οποίοι είναι σχεδόν έτοιμοι, αλλά τους λείπει το τελευταίο βήμα, θέλετε, να κάνετε το τελευταίο βήμα. Νομίζω λοιπόν ότι με τη συνδύση αυτή, με το συνδυασμό αυτό θα πετύχουμε πολύ παραπάνω αποτελέσματα στα νέα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τον ορίζοντα 2020 και σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη. Η ερώτησή μου είναι η εξής. σε ό,τι αφορά θέματα ανταγωνισμού, αλλά και την αξιοποίηση των φυτικών ταμείων για την έρευνα και την ανάπτυξη, πώς μπορούν να δημιουργηθούν τρόποι για να πετύχουμε και να συγκεντρώσουμε περαιτέρω μέσα από τον ορίζοντα 2020. Για παράδειγμα, η Πολωνία χρησιμοποιεί 20% των κοντιλίων για την έρευνα και την ανάπτυξη και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τη διάθεση των διαστατικών ταμείων για την υποστήριξη έρευνας και ανάπτυξης και το βαθμό στον οποίο λαμβάνει χρήματα ορίζοντας 2020 για το, την κλίμακα προς την αριστεία αυτή. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε και όλα τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να, ε, για όλα αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν διατυπωθεί προτάσεις μέχρι τέλη του μήνα. Μα λείπουν συγκεκριμένε προτάσει. Δυστυχώ. Ακούσαμε κάποια πράγματα για την αδελφοποίηση, το twinning, και το συνδυασμό ε, μέσων από τα δύο ταμεία, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία μπορούμε να συνδέσουμε ε, τα δύο ταμεία με τον ορίζοντα 2020. Θα δώσω το λόγο στους επιρρογνωμονές μας για να απαντήσουν. καθηγητής Γκουλίνσκι, καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τις ε, ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Να πω καταρχάς ότι αυτό που λένε οι συνάδελφοι δείχνει ότι υπάρχει πλέον κάποια συνέργεια μεταξύ των διευθυντικών ταμείων και του 7ου πρόγραμματος πλαισίου. Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι υπάρχουν φραγμοί, υπάρχουν εμπόδια παραδείγματος χάρη για τη δημιουργία περιφερειακών ε, κέντρων αριστείας ή περιφερειακών στρατηγικών. Στην Ανατολική Γερμανία, για παράδειγμα, στην Πολωνία, φαίνεται ότι ήταν πιο εύκολο να απορροφηθούν ε, οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων, άρα υπήρχαν κάποιες συνέργειες. Τα διαρθρωτικά ταμεία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία υποδομών και για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Και όταν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό ικανό, φυσικά και μπορεί κανεί ε, να υποβάλει υποψηφιότητα για προγράμματα στο πλαίσιο παραδείγματο του ορίζοντα 2020. Υπάρχει συνέργεια, θα συνεχίσει να υπάρχει φαντάζομαι και στο μέλλον, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με την ε, δήλωση ότι δεν υπήρξαν ε, εμπόδια γιατί υπήρχε η συνέργεια. Όχι. Αυτό το ένα δεν αποκλεί το άλλο και νομίζω ότι στη δική μου παρουσίαση κατέστησα σαφές ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν ε, και περαιτέρω μηχανισμοί και οικονομικής διευκόλυνσης, μεταξύ άλλων, για να προσφερθούν περισσότερες ευκαιρίες σε όσες χώρες χρειάζεται να γεφυρώσουν ακόμη το χάσμα και για να έχουμε έτσι έναν εναρμονισμένο ε, χώρο έρευνας. Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη ευφυή εξειδίκευση, πραγματικά αυτό αποτελεί ευκαιρία για τις περιφέρειες και ιδίως για όσε ε, περιφέρειες δημιουργούν κάποιες στρατηγικές εφιούς ανάπτυξης. Είναι καλό να υπάρξει ε, και εκπλήρωση των, εξάντε, των κριτηρίων εξάντε για την απορρόφηση. για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον ενιαίο, τον ευρωπαϊκό ε, ενιαίο χώρο έρευνα. Σε ό,τι αφορά υπερεθνικέ διακρατικέ πρωτοβουλίε, αυτή είναι μια καλή ιδέα γιατί μπορεί να δώσει τη δυνατότητα της δημιουργίας ε, μια ε, συνεργασίας διαφόρων περιφερειών ε, που θα δημιουργήσουν έτσι κάποια διακρατικά προγράμματα με τη συμμετοχή περισσότερων της μιας χωρών. Σε ό,τι αφορά την εδραίωση παγίωση κάποιων διεθνών κλάστερ, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε λέγοντας ότι η κακή διαχείριση ήταν το μόνο πρόβλημα σε κάποιες χώρες. Σε κάποια ερευνητικά κλάστερ και οι υποδομές αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι σημαντικά στοιχεία. Είναι απαραίτητα, παραδείγματο χάρη, τα, ε, είναι απαραίτητε οι διοικητικέ, διευθυντικέ δεξιότητε ό,τι αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο. Χρειάζονται όμως και πόροι. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί αναφέρατε την Πολωνία. Ως μια χώρα που έχει αξιοποιήσει σημαντικά τους πόρους για την έρευνα και την ε, καινοτομία. Πράγματι ε, έχουμε ήδη κάνει πρόοδο αλλά και πρέπει ακόμη περισσότερο να προωθήσουμε τα πράγματα. Παρακαλώ. Ποιος θέλει το λόγο? Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, δηλαδή να επενδύουμε τις δυνατότητες, στις δυνατότητες. Αυτό που έγινε στο Μαγδεμβούργο και στο Σουόνσι ε, μοιάζουν αυτά που, που έχουν γίνει. Είχαμε έρευνα, μετά επενδύσαμε στα διαθετικά ταμεία, μπορέσαμε έτσι να κάνουμε περισσότερο έρευνα γιατί προσέλκυσε αυτό περισσότερο κόσμο. Έτσι είχαμε λοιπόν ε, προσθετικό αποτέλεσμα. Έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο κάποιες προσπάθειες μετατόπισης κέντρων αριστείας σε κλάστερ, ομαδοποίησή του, αλλά αυτέ οι προσπάθειε απέτυχαν ε, εν γέννη, διότι υπήρχαν ε, κάποιοι οι οποίοι δεν ήθελαν να μετακινηθούν. Υπήρξαν επίσης επενδύσεις σε υποδομές που δεν βασίζονται στην αριστεία της έρευνας και έχουν μείνει πλέον κενά, κενές αυτές οι προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να έχουμε πρόσβαση μεν στην έρευνα, αλλά να στηρίξουμε την έρευνα με διδροτικά κονδύλια και μετά να δώσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας κλάστερ με εξάπλωση, διεύρυνση. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να σχολιάσει. Η κυρία Βόλφ. Να πω και εγώ δύο λόγια αν θέλετε για το θέμα του ανταγωνισμού, του οποίο ανέφερε ο κύριος Γκλάντε. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για αριστεία στην έρευνα, δεν γίνεται να, μιλάμε, να μην μιλάμε για ανταγωνισμό, αλλά θα πρέπει να βρούμε και ένα μηχανισμό ο οποίος θα εντάσσεται και στην, στα πλαίσια των διευθυντικών ταμείων. Για το πώς τα διευθυντικά ταμεία, ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες, μπορούν να συνδεθούν με τις προοπτικές της αριστείας αλλά μία τέτοια αίτηση θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία αληθοφανή, μία θεμητή ε, προοπτική για την επίτευξη αριστείας και πώς μετά την επίτευξη της αριστείας και μετά το πέρας της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής θα μπορεί να επιτευχθεί ο απότερος στόχος να εμπορευματοποιηθεί το προϊόν, να ενταχθεί στα πλαίσια των εθνικών προϊόντων, αλλά σε ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ανταγωνιστικότητα, ιδάλλως δεν θα υπήρχε η αριστεία. Μας διδάσκει η εμπειρία. Μια άλλη ερώτηση έγινε για τα βασικά εμπόδια. Εμείς στο Ομόσπονδο Κρατήδιο αναρωτηθήκαμε γιατί τόσο καιρό τα πηγαίναμε τόσο άσχημα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ να σας πω ότι και εγώ ήμουν καθηγήτρια που δεν έγραψα, δεν έκανα τις σχετικές αιτήσει. Να σας πω ότι στη Γερμανία, στην Ανατολική Γερμανία, τα πράγματα ήταν ίσως και υπερβολικά καλά και εύκολα. Είχαμε πάρα πολύ καλές συνθήκες και δεν είχαμε την έντονη ανάγκη να συμμετάσχουμε στα ευρωπαϊκά μέσα. Θα πρέπει λοιπόν οι επιστήμονες, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το διαπιστώσουμε, να έχουν και κίνητρα. Θα πρέπει να έχουν και το καρότο και το μαστίγιο. Και πριν από δύο χρόνια δημιουργήσαμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ανώτατων ιδρυμάτων για να μας υπενθυμίζει ακριβώς ε, ότι κοιτάξτε Χρειάζεται μεγαλύτερη ορμή. Χρειάζονται κίνητρα. Και να ε, δίνετε όθηση και σε αυτή την ε, τόλμη που χρειάζεται. Και νομίζω ότι αυτό μας έκανε να ξεπεράσουμε αυτό το κατόφλι, αν θέλετε, αυτό το εμπόδιο, προκειμένου να ξεπεράσουμε και να πετύχουμε κάτι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τρίτο θέμα, ο κύριος Έλλερ μας ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα. Εμείς επανειλημμένα χρησιμοποίησαμε διαφορετικά ταμεία για να ε, υποστηρίξουμε ε, έργα υποδομής το ανέφερε και ο συνάδελφος ε, στην έρευνα πάντα χρειαζόμαστε άριστους επιστήμονες όχι απαραίτητα βραβευμένους με βραβείο Νόμπελ αλλά που μπορούν να καταλάβουν τι είναι το business plan, για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να είναι σε θέση να γράψουν οι ίδιοι ένα business plan, αλλά να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Και αυτές οι προσωπικότητες, όταν μπορούμε να τις εντοπίσουμε και να τις ε, προσελκύσουμε, νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή των ιδρυμάτων Max Planck και είναι πολύ καλή στρατηγική, μπορούν να αποτελέσουν, αν θέλετε, ε, το επίκεντρο και οι υποδομές μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη λήψη της απόφασης αυτής από πλευρά των επιστημόνων. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτή την προϋπόθεση μπορούμε να πετύχουμε κάτι προκειμένου να μην καταλήξουμε να έχουμε τις τέλειες υποδομές χωρίς όμως να έχουμε και τους ανάλογους επιστήμονες. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εγώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία εμπειρία από μία πορεία προς την αριστεία και επιστροφή σε τοπικό επίπεδο, κάτι που ακροθυγώς έδειξα και πριν. Το δίκτυο δημόσιων φορέων που ήδη και από το Ένστρετ. Στα πλαίσια, ξέρετε και το Φέστρετ, για τις ε, περιφέρειες σύγκλησης σε εθνικό επίπεδο για να μπορέσει να προβεί με κλιμακωτό τρόπο στην ε, καλύτερη συνάθρηση αυτών των δικτύων ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει πρωτοβουλία ΕΣΦΡΗ. Αυτές τις μέρες είχαμε τα εγγένεια κάποιων ε, από αυτά τα κέντρα σε τοπικό επίπεδο που γεννήθηκαν, επαναλαμβάνω, από την παρέμβαση έστρα. Και συνδέονται όμως ε, με κάποιες από τις πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκού Επίπεδου για την Αυτές οι υποδομές, σε αυτές μάλλον τις υποδομές, ε, προσδόθηκαν οι ικανότητες κάποιων ανώτερων ερευνητών και τίποτα δεν πρόκειται να προχωρήσει αν δεν στηριχθούμε στους ίδιους τους ανθρώπους. Αυτοί οι ερευνητές εκπώνησαν αυτή την κλιμακωτή, αν θέλετε, προσέγγιση της έρευνας από τα τοπικά εργαστήρια έως την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, έως μια περιφερειακή πρωτοβουλία που εφάρμοσε το ΕΣΝΙΠ με το όνομα Περιφερειακές Συνεργασίες για την Καινοτομία δημιούργησαν κλάστερ με επιχειρήσεις της απολίας για project έρευνας που συνδέονται και με τα θέματα που απασχολούν και όλη την Ευρώπη εν γέννη. Άρα, όπως είπα και πριν, υπάρχει δυνατότητα να κάνεις μια πορεία ξεκινώντας από τοπικό επίπεδο, να φτάσεις στην αριστεία και να επιστρέψεις πάλι στο τοπικό επίπεδο. Εγώ δεν πιστεύω στην ε, υπάρξη μόνο ενός και μόνο εργαλείου πανάκια. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ένα παζλ ε, όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν τα προγράμματα. Μια τέτοια στρατηγική εγώ πιστεύω και πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει και το εξή ζήτημα πώς θα ε, χρησιμοποιηθεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ε, αυτή η ερεύνα των προκαπαιδών. Και η δημόσια ζήτηση, η ζήτηση που υπάρχει ε, από το δημόσιο τομέα σε όλε τι περιφέρειε. είναι μια τυχελή Ευχαριστώ πολύ κύριε Κωνσταντζα Κρίλ και μετά η κυρία Μαρία Καρβάλιο. Σα ευχαριστώ Καταρχά να ευχαριστήσω του υπουργού ε, και τι υπουργού ε, για το ότι δεν χρειάζονται τόσα, πολλές, τόσα πολλά μέσα χρηματοδότηση. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε. Σύνδεση ορίζοντας 2020 και των παιδικών ταμείων που βρίσκεται. Ένα, μία από τις θεματικές προτεραιότητες, μία από τις πιο σημαντικές ε, θεματικές προτεραιότητες η έρευνα και η καινοτομία βρίσκεται στην πολιτική μας ατζέντα και τώρα στην πρότασή μας για το κοινό ε, στρατηγικό πλαίσιο κάνουμε τη σύνδεση με τον ορίζοντα 2020 και με τις συνέργειες που μπορούν να προκύψουν Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να τα εξετάσουν αυτά για να δουν κατά πόσον να πιστεύουν ότι υπάρχουν ε, στοιχεία στο κοινό στρατηγικό πλαίσιο, τα οποία ενδεχομένως μπορούμε να τα προσθέσουμε στην γενικότερη ε, προσέγγιση. Μέχρι 7 ε, Ιουνίου έχουμε χρόνο και εγώ και ο Λάμπερτ όσοι συνεισηγητές είμαστε ανεκτοί για συζήτηση για αυτό το θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Αυτό όμως που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι το εξή. Φυσικά υπάρχει αντίφαση σε ό,τι αφορά την προώθηση της αριστείας και την προώθηση ε, την ε, εγκάρσια, αν θέλετε, αλλά οι περιφέρειες ε, καλούνται να επιδείξουν τέτοια δυνατότητα καινοτομία ως όρο εξάντε και εκεί βλέπουμε ότι τα λειτουργικά προγράμματα στις περιφέρειες στο επίπεδο Υπουργείων υπάρχει επαφή με τα ιδρύματα προκειμένου να καταρτιστεί μια κοινή στρατηγική για κάθε περιφέρεια προκειμένου να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτό μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της ε, ενίσχυσης ε, της αριστείας, αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί στην ενίσχυση των ερωτικών ταμείων. Νομίζω λοιπόν έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία και αυτό θα πρέπει ουσιαστικά να αποτελεί το στόχο μας προκειμένου οι περιφέρειες να έχουν την δυνατότητα να κάνουν έρευνα αριστεία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Καρβάλιο. Very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, ο ορίζον 2020 αφορά την αριστεία. Αλλά θα πρέπει να μπορεί να καλύψει και τις ε, νεοσυστηνόμενες ε, μονάδες ε, Σημαντική είναι και η ευφύης εξειδίκευση, αλλά και στον ορίζοντα 2020 και στα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να έχουμε ε, αυτή την κλίμακα, αυτή τη σκάλα προς τον αριστεία. Θα πρέπει να γεφυρωθούν δηλαδή αυτά τα δύο. Θα πρέπει επίσης να είναι συγκεκριμένες οι δράσεις. Ακούσαμε σήμερα κάποια παραδείγματα. Θα σας δώσω και εγώ άλλα δύο παραδείγματα και θα ήθελα να στήσω την άποψή σας για αυτά. Είμαι εισηγήτρια για το ειδικό πρόγραμμα για τον ορίζοντα 2020 και μια από τις προτάσεις είναι ο ορίζονα χορηγεί μια σφραγίδα αριστεία σε διάφορες προτάσεις όπως το Marie Curie, προτάσεις ε, καλές ή άριστες που όμως δεν χρηματοδοτήθηκαν διότι υπάρχει συνήθως ε, ένα ποσοστό των προτάσεων που χρηματοδοτούνται. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει μια ταχεία διαδικασία ή αν δια υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια και είναι προτεραιότητα να μπορούν να χρηματοδοτούνται για τις περιφέρειες και από τις περιφέρειες κάποια προγράμματα. Δεύτερον, ο Ορίζον 2020 καλύπτει πλέον και την καινοτομία, όλη την αλυσίδα. Έχουμε λοιπόν και τα πιλωτικά προγράμματα και την επίδειξη. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθούν τα πάντα από τον Ορίζοντα 2020. Άρα η πολλαπλή χρηματοδότηση, το λεγόμενο multi-fund approach, είναι μια καλή προσέγγιση που όμως πρέπει να λειτουργήσει με απλό τρόπο. Πώς μπορούμε δηλαδή να συγχρηματοδοτήσουμε μεγάλα προγράμματα επίδειξης, βιομηχανικής επίδειξης και από τα διορθωτικά ταμεία με έναν απλό τρόπο και φιλικό προς τον ενδιαφερόμενο. Και μια άλλη υπόδειξη τελευταία κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για απλούστευση στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020 και κάτι αντίστοιχο πιστεύω πρέπει να γίνει και για τα διαρθρωτικά ταμεία. Γιατί αν υπάρχει γραφειοκρατία και αν είναι πάρα πολύ πολύπλοκα αυτά τα ζητήματα, ιδίω αν υπάρχει συνέργεια, πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Δεν θα είναι εύκολη συνέργεια. Ο πρόεδρος Μπούζεκ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, όπως είπατε, ε, υπάρχει ήδη κάποια ε, συνεργασία. Ε, ήδη πριν από έξι χρόνια με την Επίτροπο τότε Χούμπνερ και τον Επίτροπο Ποτότσινγκ που είχαμε πει τότε ότι ήταν απαραίτητη η συνεργασία αυτή. Και κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Βέβαια, ίσως δεν ήταν αρκετό το βήμα από την πλευρά δηλαδή, της περιφερειακής ανάπτυξης και από την πλευρά της πολιτικής για την ανάπτυξη και την, ε, για την έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να σας πω ότι γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, στα ταμεία αυτά. Το πρώτο προκαθορίζεται γεωγραφικός, η κατανομή έχει να κάνει με την τοποθεσία, με το χώρο και το δεύτερο όχι, δεν ε, καθορίζεται γεωγραφικά. Δεν υπάρχει γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων. Θέλω να πω το εξή λοιπόν. Ουσιαστικά εξαρτάται από την απόφαση που θα λάβουν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες εν τέλει, αν δηλαδή θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους ε, πόρους ε, σε αυτή την κατεύθυνση που εμείς προτείνουμε. Εμείς μπορούμε να απευθυνθούμε μόνο ε, στους εκπροσώπους των κρατών μελών, έχουμε κάποιου από αυτού εδώ, αλλά και στι περιφέρειες. Να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυνατότητα αυτή. Τελείως διαφορετική κατάσταση είναι αυτή που ισχύει για τον ορίζοντα 2020. Φυσικά και δεν εστεύτηκαν με απόλυτη επιτυχία οι προσπάθειες στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου. Και γιατί. Γιατί δεν είχαμε παρκή ε, συμμετοχή, για παράδειγμα, τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα ή δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο του 7ου προγράμματο πλαισίου. Σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε στην αριστεία αλλά πρέπει να γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι πολύ πιο δύσκολη η καιρή πριν, σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από 6-7 χρόνια. Πώς ε, ε, να μην είναι σημαντικό ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ταλέντα, να ανακαλύψουμε ταλέντα σε όλη την Ευρώπη. Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να βελτιώσουμε το πρόγραμμα Horizon 2020 αλλά δεν θα πρέπει ε, να χάσουμε την εστίαση, να μην βγει από το επίκεντρο η αριστεία. Αυτό είναι προφανές. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση στις ε, ερευνητικές υποδομές αριστείας. Η κυρία Καρβάλιο μίλησε και για την απλούστευση, ανάγκη απλούστευσης και στις δύο περιπτώσεις. Πράγματι, επίσης μικρομεσαία project, μικρομεσαία έργα. Σημαντικό. Μην χάσουμε την αριστεία βέβαια, αλλά ίσως θα ήταν πιο εύκολο σε ομάδες ε, από περιφέρειες συνοχής να ξεκινήσουν τέτοια ε, project. Αυτή επίσης η έννοια της ε, εφιούς εξειδίκευσης θα μπορούσε και αυτή να αξιοποιηθεί με πολύ καλό τρόπο. Και τώρα ένα άλλο παλιό πρόβλημα που υπάρχει των σημαντικών διαφορών στους μισθούς των ερευνητών. Πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό το παλιό πρόβλημα Θέτω το ερώτημα, ε, είναι δύσκολο, αλλά είναι και ε, ένα αγκάθι, αν θέλετε, στη συνεργασία μας. Πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά. Πρώτα απ' όλα για τον ορίζοντα 2020, γιατί τα πάντα εξαρτώνται από την απόφαση που θα ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό, από το Κοινοβούλιο και σε σχέση με όλα τα προγράμματα αριστείας. Εγώ θέλω να απευθύνω την εξής έκκληση. Ας κάνουμε όλες τις δυνατές αλλαγές στο πρόγραμμα Horizon 2020 προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς όμως να πάψουμε να εστιάζουμε στην αριστεία. Ευχαριστώ πολύ. Πολλοί εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δύο είναι σίγουρα που έχουν το ρόλο του Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον Γιάνν Σμιτ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά αν θέλετε για κανένα δίλεπτο να πείτε τη γνώμη σας. Thank you very much. Well, not that desperate, but that... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν είναι ότι πιέζουμε πάρα πολύ να πάρω το λόγο, αλλά μια και μου το δίνετε, να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσε και οι περιουσιάσει ε, και η συζήτηση. Τρία πράγματα έμαθα από τη συζήτηση. Πρώτον, θα πρέπει να σεβαστούμε το γεγονό ότι τα εργαλεία, τριωτικοταμεία και πρόγραμμα πλαίσιο έχουν διαφορετικού στόχου. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίω ότι οι στόχοι ε, έρχονται σε σύγκρουση μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα, αλλά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα διαφορετικά μια είναι η δημιουργία δυναμικού, εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων, νέο εξοπλισμό, δημιουργία τοπικών επιχειρήσεων. Ο ρόλο του ορίου 2020 είναι να συνδέσει την αριστεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, το πρώτο που έμαθα από τι μέρε παρουσιάσει είναι ότι τα εργαλεία αυτά έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν θα πρέπει να συγχωνευτούν, αλλά να έχουν στενή συνεργασία. Το δεύτερο και σημαντικό που έμαθα σήμερα είναι ότι, όπω είπε ο κύριο Μπούζεκ, είναι πολύ σημαντικό οι περιφέρειες να εκπονήσουν μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Αν δεν υπάρχει αυτή η στρατηγική, δεν υπάρχει κλίμακα προς την αριστεία. Άρα όσοι τρέφουν τη φιλοδοξία να ανέβουν αυτή τη σκάλα της αριστείας, είδαμε και το παράδειγμα της ε, απουλίας, ακριβώς αυτό μας δίδαξε. Και το τρίτο που έμαθα σήμερα είναι η αναγκαιότητα να υπάρξει πολύ καλή διασύνδεση των διαφόρων εργαλείων. Οι κανόνε τη χρηματοδότηση και δικασία να είναι τέτοιε ώστε στο τέλο ε, το ποθητό να ε, δίνει αποτελέσματα και όχι το αντίθετο. Θα πρέπει λοιπόν και εσείς στο Κοινοβούλιο και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν να υπάρχει αυτή ε, η διασύνδεση για να μπορούμε να επιτύχουμε τις συνέργειες στη συμπληρωματικότητα. Τέλος και σημαντικό, χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί δεν έγινε αναφορά στην διαφορά ανάμεσα στις χώρες της διεύρυνσης και τα παλιά κράτη-μέλη. Ακόμα και στη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ιταλία υπάρχει ζήτημα αριστείας. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, σαφής ε, ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα τα νέα κράτη-μέλη της διεύρυνσης και τα παλαιά. Όλοι έχουν ανάγκες, οπότε είναι καλό να μην θέτουμε τη συζήτηση υπ' αυτό το πρίσμα. Δεν είναι κάποια κράτη-μέλη αντί κάποιον άλλον, είναι κάτι που μας απασχολεί όλους και πρέπει να το Ευχαριστώ πάρα πολύ και ο κύριος Μάρτιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την ε, οργάνωση αυτή της ακρόασης ε, και για τους τέσσερις αγορητές ήταν πραγματικά πολύ διαφωστικές τις παρουσιάσεις γιατί μιλάμε για αφηρημένες έννοιες πολύ συχνά αλλά να έχουμε αυτά τα παραδείγματα πάρα πολύ καλό και κρίσιμα είμαστε, γιατί ήδη για την κείμενη δημοσιονομική περίοδο βλέπουμε ότι ένα τέταρτο περίπου τη κοινωνική μορτοδότηση πάει στην έρευνα καινοτομία. Μιλάμε για κάτι τετραπλάσιο σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και θέλουμε και υψηλότερο ε, ποστό να επιτύχουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Γι' αυτό, όπω είπε ε, κύριε Κρέλ, η έρευνα και η καινοτομία είναι ένα στους βασικούς και πρώτους στόχους χρηματοδότησης και συνδέεται με τα ελάχιστα ποσοστά της χρηματοδότησης, βεβαίως για να υπάρξει σωστή εστίαση της χρήσης του Ταμείου ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξουν αυτές οι συνέργειες και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συνέργειες. Όπως είπε ο Ρόμπερτ Γιάννης βεβαίως, το σημαντικό είναι να μετατρέψεις τις ιδέες σε κάτι ε, απτό και λειτουργικό. Δεν είναι κάτι καινούργιο για την προγραμματική περίοδο, αλλά γίνεται όλο και πιο σημαντικό με βάση τη θέσιμα κονδύλια. Οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε με σαφείς έννοιες. Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια ιδεών και ενιών. Βλέπουμε ότι ο ορίζοντας 2020 εστιάζει στην αριστεία και από εκεί και πέρα έχουμε την χρηματοδότηση του Περιφερειακού Ταμείου ε, που βλέπει την ένωση τοπικό επίπεδο, ενίσχυση της έρευνα και της οικοδόμησης δυναμικού από την άλλη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς της γνώσης των αποτελεσμάτων της έρευνας επίσης. Από τις παρουσιάσεις που είδαμε σήμερα, ε, είναι σαφής σε διαφοράς επιδονιών, αλλά υπάρχει η συμπληρωματικότητα. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε εναρμονισμένους κανόνες και στο τομέα στον οποίο έχουμε κάνει πρόοδο. Αν δείτε την πρόταση Κομισιόν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και βλέπετε σημερινή πρόταση, βλέπετε ότι ε, καταλήγουμε σε μια κοινή δέσμη κανόνων επιλεξιμότητας που πλέον δεν αποτελούν πρόσκομα στην όλη προσπάθεια. Έπειτα άλλα ε, προβλήματα όπως ε, είναι τα ε, καταποκοπήν δαπάνες, το ΦΠΑ, η χρήση άλλων εργαλείων από άλλους τομείς πολιτικής κλπ. Είναι όλα πράγματα που λαμβάνουν υπόψη. Έπειτα, πώς μπορεί όλα αυτά να είναι λειτουργικά σε επίπεδο κρατών μελών, σε επίπεδο Περιφερειακού Ταμείου και Ταμείου Συνοχής. Θεμελιώδους σημασία αυτό γιατί εδώ μετουσιώνονται οι ιδέες στην πραγματικότητα. Και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι, χρειάζεται, ότι πρέπει να έχουμε αυτή τη στρατηγική που θα μας επιτρέψει όλες τις ιδέες ε, να τις κάνουμε πράξη με την καλύτερη δυνατή χρήση ε, των κονδυλίων. Εκεί εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη να τα κάνουν αυτά πράξη. Ε, μέσα, στα, μέσα στα πλαίσια της πλατφόρμας της Εβίλης που αναφέρθηκε και νωρίτερα. Και τέλος, αυτό που πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε είναι ότι έχουν λάβει όλα τα δεδομένα οι δικαιούχοι. Ήδη έχουμε κάνει έναν οδηγό για τους δικαιούχους που έχει επικαιροποιηθεί, που τους ενημερώνει για τις διάφορες πηγές χρηματοδότηση και τους τρόπους πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Έχουμε μια νέα λοιπόν εκδοχή θα έχουμε μάλλον μια νέα εκδοχή αυτού του οδηγού όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει για την νέα δημοσιονομική περίοδο. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε παρά τι προσπάθειε που κάνουμε ε, είναι εξή. Έχουμε δύο διαφορετικά εργαλεία χρηματοδότηση. Στο ένα εργαλείο έχουν ε, κοινή, αν θέλετε, αρμοδιότητα διαχείριση στα κράτη-μέλη, ενώ στο άλλο εργαλείο έχουμε μια κοινή συγκεντρωτική, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαχείριση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κατάλληλη συνεκτικότητα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε του ε, στόχους. Και να γεφυρώσουμε αν θέλετε κάποια στοιχεία μεταξύ των δύο εργαλείων και αυτό θα γίνει με τις ε, συμφωνίες σχέσεις, ώστε οι συνέργειες που λέμε και ξαναλέμε να γίνουν πράξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκολας. Και η τελευταία κουβέντα ανήκει στους προσκεκλισμένους μας. Ποιοι επιθυμούν να πάρουν το λόγο, παρακαλώ. Δεν σας αναγκάζουμε αν το επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Εν συντομία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε δύο πτυχές για την ιδέα της ε, ανάπτυξης μέσω της ε, ε, γνώσης, τη διαχώρηση, τη διάκριση μεταξύ της εφεύρεσης και της καινοτομίας. Δηλαδή υπάρχει ένας τομίας που περιλαμβάνει την διάδοση της γνώσης, τη μεταφορά της γνώσης. Δεν ε, συμπεριλαμβάνει απαραίτητα, ξέρετε, ε, βραβευμένους με Νόμπελ. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορεί να αξίζουν τον κόπο χωρίς να είναι ε, προγράμματα εχμής. Αυτά εντάσσονται στην ορίζοντα 2020. Κάτι δηλαδή που μπορεί να μην είναι ανταγωνιστικό, αλλά που μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη μιας κάποιας περιφέρειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κανείς άλλος, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να πούμε με σαφήνεια ότι και το Horizon 2020 και τα δραστηριοτικα ταμεια Ταμεία 2014-2020 δίνουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες για τις χώρες οι οποίες ακόμα προσπαθούν να φτάσουν σε ένα κάποιο επίπεδο και ότι πολλά εξαρτώνται από αυτές τις χώρες. Λοιπόν, θα ήθελα να υπάρξουν απλουστεύσεις σε ό,τι αφορά τη συνέργεια μεταξύ των δύο προγραμμάτων για να ωφεληθεί όλη η επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Καρβάλιο. Αυτό που για πρώτη φορά εμφανίζεται είναι το Marie Curie, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν θύλακες αριστείας σε όλη την Ευρώπη και θέλουμε ανταλλαγή φοιτητών και αυτό θα ωφελούσε τους πάντες. Υποστηρίζουμε όλα όσα είπε από πλευράς πρακτικής ε, σε ό,τι αφορά την υποβολή αιτήσεων και για να σχολιάσω αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητήριος δύναμη θα είναι οι τομείς όπου, χρειάζεται, ε, όπου υπάρχει φιλοδοξία και μετά χρειάζεται στρατηγική για την ανάπτυξή της. Ναι, σε ό,τι αφορά τα θέματα εξειδικευσής και πώς ε, την πετυχαίνουμε, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι πρόκειται για έναν δρόμο που τους πρώτους μήνες του 2013 δεν θα μας οδηγήσει μόνο να αυξήσουμε τα τριφωτικά ταμεία. Προτάθηκε να χρησιμοποιήσουμε τον δρόμο αυτό για να καταδείξουμε τι μπορεί να οδηγήσει σε αριστεία, που υπάρχουν περιφερειακοί φορείς οι οποίοι μπορεί να το πετύχουν αυτό σε συνεργασία με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Και αυτό έχει να κάνει και με την ανάγκη των περιφερειακών φορέων σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και της συνολικής περιφέρειας. Να χρηματοδοτηθούν τέτοια έργα έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με διάφορες προσεγγίσεις που περνάνε μέσα από τα περιφερειακά ταμεία. Αυτό αποτελεί ασφαλώς ε, προϋπόθεση και δεν είναι τυχαίο ότι στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο υπάρχει έρευνα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη χρήση του υδρογόνου. Χρειάζεται μια απλοποίηση των ε, νομοθεσιών. Αυτό σίγουρα είναι επιθυμητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται η ακρόαση μας, λέει η Πρόεδρο. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή. Η Επιτροπή Ρέτζι παρακαλώ να παραμείνει στην αίθουσα. Όλοι οι υπόλοιποι, αν θα θέλετε να αποχωρήσετε, γιατί έχουμε ψηφοφορίες. Dear colleagues, we have a lot of... Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μία μακρά και δύσκολη σειρά ψηφοφοριών. I, I am going to check whether your machines were... Να ελέγξουμε πρώτα απ' όλα αν δουλεύουν τα μηχανήματά σας, για αυτό σας παρακαλώ να εισάγετε τις κάρτες σας. η αριστεία ας μείνει η σκάλα να φύγει, το stairway. Could you, can, can we check the vote? Can we open the... Παρακαλώ να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Υπάρχουν δύο οι οποίοι έχουν ε, βάλει τις κάρτες μένα, αλλά δεν έχουν ψηφίσει. Τέλο πάντων, για του περισσότερου φαίνεται ότι λειτουργεί. το μηχάνημα και γι' αυτό, ναι, Κωνσταντσε. Ντανούτα, μία έκκληση. Στην πρώτη γνωμοδότηση έχουμε μία σειρά τροπολογιών για τις οποίες δεν είμαστε αρμόδιοι, γιατί αναφέρεται, για παράδειγμα, τροπολογία 66, 74, 75, ότι αυτό μπορεί να υπερβαίνει την αρμοδιότητα της ΡΕΓΚΙ ε, να μην ψηφίσουμε καν τότε στην περίπτωση αυτή. Αυτό θα ζητούσα. So there is a proposal coming. Υπάρχει λοιπόν πρόταση από τους σοσιαλιστές για όσα θέματα δεν άπτονται τη δική μας αρμοδιότητα να μην ψηφίσουμε. Αν κατάλαβα καλά, είναι κάποιος αντίθετος σε αυτή την πρόταση. Για τις, μιλάμε για τις τροπολογίες στην έκθεση Πιότερ Πορέμπα. Τροπολογίες ποιες, 66. Α, πολλές είναι. Άρα θα τις παρακάμπτω στην ψηφοφορία, αν συμφωνείτε. Κύριε Πορέμπα, συμφωνείτε. Και ο Λάμπερτ βλέπω ότι συμφωνεί, άρα υπάρχει πλειοψηφία. Λοιπόν, ξεκινάμε την ψηφοφορία για την έκθεση Πορέμπα. Τροπολογία 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 54. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται αν δεν κλάψουν οι σοσιαλιστές θα θεωρήσουμε ότι απορρίπτεται. 55 υπέρ. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. 55 κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 56 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την τροπολογία 56 άρχεται η ψηφοφορία. It's rejected. Απορρίπτεται. Με μικρή διαφορά, αλλά απορρίπτεται παρόλα αυτά. 21 ψήφοι κατά 19 υπέρ. Λοιπόν, 57 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές. Εδώ δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, άρα ελέγχουμε την 57. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά... Πέραση ψηφοφορίας, πράγματι εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι καλό θα ήταν να ελέγξουμε την 60 γρήγορα γρήγορα άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται τροπολογία 61 υπέρ κατά Το ίδιο. Να ελέγξουμε την 61. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Ψήφι υπέρ. 62. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απο... μάλλον να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 64, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 25 ήταν η ψήφη κατά. 65 εγκρίνεται, 67 υπέρ, κατά, Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ε, μπορώ να καταλάβω, να ελέγξουμε την 67. Μάλιστα, οπότε βλέπω ότι έχουμε τις ίδιες ε, συμμαχίες συνασπισμούς, άρα δεν θα ελέγχω από εδώ και πέρα. 68 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά Ελέγχουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με την ίδια διαφορά. 71 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 9 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 73 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται Πάμε στη 10 τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Όχι. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 όχι που πάμε 87 υπέρ κατά να ελέγξουμε τα 87 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε και τη 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Υπάρχει προφορική τροπολογία που αντικαστά το older από το elderly. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Τη 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Ναι, ωραία. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 104. Όχι. 105 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 106. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 100. 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 109. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε την 109. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 110. 110. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 111 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 112 όχι. 116 αγαπητοί συνάδελφοι ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 19 καταπίπτει. 118 ψήφι υπέρ, Κατά αποχές εγκρίνεται. 119 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. 121 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε τον 127. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 128 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. είναι διερεμένη σε ομάδες αγαπητοί συνάδελφοι. Ξαναρωτώ, ψήφι υπέρ της, της 21, της 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε σε τελικές σκέψεις. 23 τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, ελέγχουμε την 24, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 ψήφι υπέρ. Υπάρχει προφορική τροπολογία, Λάμπερτ. Είναι γλωσσική η τροπολογία. Την κυρία Κράτσα προέρχεται, ναι. Θέλετε να την παρουσιάσετε ή να το κάνω εγώ. Στο μικρόφωνο παρακαλώ. Union and its regions. I propose. Yes. So the text, the, te the original text. text. The original text. I don't have the original text. Yeah. Δηλαδή το πρωτότυπο. Ναι, το έχω εγώ και λέει. Time of economic crisis in the EU as a whole and in individual regions. And the new text is... Και το νέο ε, κείμενο λέει ότι σε αυτές τις ε, περιοχές, σε αυτή την εποχή κρίσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ε, περιφερειές της. Μάλιστα. Ωραία. Βελτίωση λοιπόν Ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική 2, δεν πιστεύω ότι είναι κανείς κατά. Λοιπόν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ. Να σηκώνετε τα χέρια σας κατά αποχές. Να ελέγξουμε την τροπολογία 1. Closed. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε την τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 37. Είναι μια ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές νομίζω εγκρίνεται. Δεν συμφωνείτε. Να ελέγξουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Το ΕΛΚ ε, θεωρεί ότι αφού αυτό δεν είναι υπέρ, δεν εγκρίνεται και τροπολογία. Και έχουν και δίκιο. Το δεύτερο τμήμα συγκεκριμένα. Λοιπόν, τροπολογία 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 40 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 41 κατά τμήματα, αλλά θα ψηφίσουμε μόνο το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ. Κατά Αποχές. Ξανά. Ποιοι είναι υπέρ 43. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε, εντάξει. Είδατε πώς σας ξυπνάω. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 παρακαλώ θέλετε το λόγο. Τη 41, το δεύτερο τμήμα, αν δεν απατώμε, δεν το ψηφίσαμε. Το ψηφίσαμε και απορρίφθηκε. Α, όχι, έχετε δίκιο. Το πρώτο να ψηφίσαμε, γιατί το δεύτερο καταπίπτει. Τη 48 ψηφίζουμε τώρα. Ψήφι υπέρ, 48. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται νομίζω. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία Uh, Θα πρέπει να ψηφίσουμε για την ε, γνωμοδότηση συνολικά. Έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία. Δεν έχουν ψηφίσει όλοι. Τώρα σχεδόν όλοι έχουν ψηφίσει. Λοιπόν, εγκρίνεται 39 ψήφοι υπέρ. Συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία έκθεση Ολενίτσακ. Και πάλι πρόκειται για μια μακρά και δύσκολη ψηφοφορία. I have Άρχεται ψηφοφορία, αγαπητέ συνάδελφοι. Είπαμε τροπολογία 49. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα υπάρχει μία πρόταση να ψηφίσουμε ομαδικά τις τροπολογίες 52-60. 52 έως και 60 μπορούμε να ψηφίσουμε ομαδικά. Όχι. 52-59 ούτε. Οι πράσινοι λένε όχι. Λοιπόν, χάνουμε το χρόνο μας. 52 υπέρ. Κατά. Μην το ξεχνάτε, λέει η πρόεδρος. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 Συγγνώμη, πέρασα την 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η Κωνσταντσα συνεχώς είχε το χέρι της ψηλά και είχα μπερδευτεί. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίφεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίφεται. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται μου λέει ο βοηθός. Ελπίζω να είναι σωστό. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείται. Συμβασμό 2 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβασμό 3 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. υπάρχει μια πρόταση για να ψηφίσουμε τις 74 έως 87 ομαδικά. Ναι, ωραία, ευχαριστώ. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της ομάδας τροπολογικών 74 έως 87, υπέρ κατά αποχές εγκρίνοντα. Πάμε στην 88. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 4 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 92 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 95 δεύτερο, συγγνώμη, το πρώτο μέρος μόνο ψηφίζουμε. 95 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ. Όχι, έχω κάνει λάθος. Καταπίπτει. 110 καταπίπτει. Λοιπόν, έχει γίνει μια αλλαγή στον κατάλογο ψηφοφορία την τελευταία στιγμή και μου λένε ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Αν δεν ψηφίσαμε θα διαγραφούν. Λοιπόν, 110 ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, Αποχέ, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείτε. 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 117. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 120 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 121 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 122 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 16 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 17 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 129 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 130 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται 131 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται 132 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται 134 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 137 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 139 υπέρ, με συγχωρείτε. 139. Δυσκολεύουμε, δυσκολεύουμε αυτό το κατάλογο, λέει ο Πρόεδρος. Προφορική τροπολογία. Κανεί δεν είναι κατά της τροπολογία, άρα ψηφίζουμε την 139 όπω τροποποιήθηκε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 8. Υπέρ. Κατά αποχές Υιοθετείτε. 142. Ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 23. Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 147 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 148 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω είναι 148 ελέγχουμε Α, ε, ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται 152 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται 25 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται 153 Σωστά. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές Υιοθετείται 160 υπέρ. Κατά υποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Έτσι μου φαίνεται. Ελέγχουμε την 160... Όχι, όχι. Την 161 λέει η πρόεδρος. Check on 160. Okay. Ελέγχουμε την 160. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Είδατε πόσο το είπα. 161 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 164 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 165 υπέρ Θέλετε να ελέγξουμε την 164. Ελέγχουμε την 164. Check Πέρας υιοθετείτε, όπως είχα πει. 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 166 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 26 συγγνώμη 170 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 171 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 172 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 173 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 27 Ποιος είναι υπέρ της 27, ποιος είναι κατά. Είσαστε και υπέρ και κατά, συνάδελφε. Για να ελέγξουμε την 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Colleagues 27 Συνάδελφοι, την 27, ηλεκτρονικός έλεγχος. Adopted I made a mistake, Να, έκανα λάθος. Υιοθετείτε, πάντως. 28. Ποιος είναι υπέρ? Για την 28 ψηφίζουμε. Κατά, αποχές. Υιοθετείτε. 29, υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε 30 υπέρ. Παρακαλώ, για 30 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείτε ή όχι. Να ελέγξουμε την 30, ελέγχουμε την 30. Yeah, because I'm... we vote. Άρχεται ψηφοφορία για την 30 την 30. It's very slowly. You, you are voting very slowly because... Ψηφίστε πάρα πολύ αργά, συνάδελφοί μου. Βλέπω τόσο κόσμο που και δεν ψηφίζει. Δέκα ακόμη δεν έχουν ψηφίσει. Την 30 ψηφίζουμε, συνάδελφοι. Απίστευτο είναι. Δεν μπορούμε να κλείσουμε άμα δεν έχετε ψηφίσει. Λοιπόν, κλείνω, κλείνω την ψηφοφορία. Και απορρίπτεται. 31 υπέρ. Όχι, τέλειωσε η ψηφοφορία. Λοιπόν, κατά αποχές υιοθετείτε. Η 32 υπέρ κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Δεν σηκώνω τα χέρια σας. Απλά φαντάζομαι το καθένα ψηφίσει ανάλογα με τη γραμμή τη ομάδα, έτσι. Μια χαρά κάνετε. Ό,τι λέει ο Λαμπέρ να κάνετε, αλλά. Λοιπόν, την 32. Υπέρ. Κατά. Είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, ελέγχουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Open. Άρχεται η ψηφοφορία. Close the Υιοθετείτε 33 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 34. Ελέγχουμε την 33. And Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Πάμε στα εκτιμώντα Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές υφετείται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 42 ο Λαμπέρ ψηφίζει έτσι λοιπόν ε, κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 2 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 44 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 45 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε τη 45 άρχεται η ψηφοφορία ελέγχουμε τη 45 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τελική ψήφο ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. η ψηφοφορία. Να σας ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε. Ναι, βεβαίω. Για το άρθρο, μισό λεπτό να το βρω. Παράρτημα 2, παράγραφος 1, 139, ανανεώσιμα συστήματα αντλησής για την εκμετάλλευση της ανανεώσιμης ενέργειας. Αν σωστά γνωρίζω, η μοναδική κατάσταση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντλήσεις αντλίες για την ε, αποθήκευση ενέργειας είναι και τη γεωθερμική ενέργεια, για την ηλιακή ενέργεια και για την αιωλική ενέργεια δεν χρησιμοποιούνται αντλίες. Για τη μοναδική ενέργεια που χρησιμοποιούνται αντλίες. Ναι, ναι, ναι, μα γι' αυτό το απορρίψαμε, λέει η Πρόεδρος, γιατί το ξέρουμε ότι δεν βγάζει νόημα. Α, πολύ ωραία. Εντάξει. Can you Can you allow me to vote? Ναι, επιτρέψτε μου να ψηφίσω. Κάποιος μου κλείσε το μηχάνημα και δεν μπορώ να ψηφίσω. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος και περνάμε έτσι στην έκθεση Λουκατσιεύσκα. Στο 7 στη σημερινή διαταξή. Θα ψηφίσουμε γνωμοδότηση για το μηχανισμό πρωτεξιατικής βοήθειας, που είναι και πιο σύντομος. Να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 4, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 24. Με προφορική τροπολογία δεν ξέρω αν είναι κανεί κατά. Όχι, εντάξει, να το ψηφίσουμε από τροποποιείται. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26. Υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. 9. Υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 10. Υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 27. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές. Α, δεν ξέρω να το ελέγξουμε. Αν θέλετε πρώτο τμήμα της 27. Closed and it's, uh, it's adopted. 21 to 20. Μάλιστα, λοιπόν, το ενεργειακό το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 28, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται και πάμε στις τελικές σκέψεις. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ. Κατά δεν ξέρω να το ελέγξουμε. Για την 14 παρακαλώ. Ελέγχουμε το 14 έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Α, καταπίπτει. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου έκθεσης, γνωμοδότησης, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Πολύ ωραία, εγκρίνεται, συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στην έκθεση του Γιώχιμ Τσέλερ για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας. Αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ, κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται 24, αλλά στο ελέγξουμε αν θέλετε. Αλλά μου φάνηκε ότι εγκρίνεται. Ψηφίστε παρακαλώ για να κλείσει η ψηφοφορία. Ωραία. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 με προφορική τροπολογία αν δεν είναι κανεί κατά να ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 α, 32 υπέρ κατά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 Έναρξη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν ε, κατάλαβα αν θέλετε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε την 46. Έναρξη και πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ. Κατά με προφορική τροπολογία στην 49 να ψηφίσουμε όπως έχει τροποποιηθεί. Να ελέγξουμε λοιπόν την ψηφοφορία για την 49 ηλεκτρονικά. Έναρξη και πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται η 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στα ιστολογικές σκέψεις συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο 26 έχουμε μία προφορική τροπολογία υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Περνάμε στο τελευταίο λοιπόν θέμα. Τελευταία ψηφοφορία. Εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον υπολογισμό 2013 Γιώργος Στραφωτικάκης. Τέσσερις τροπολογίες. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται τελική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Πάρα πολύ ωραία, εγκρίνεται. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τις ε, ψηφοφορίες μας και ας περάσουμε να δώσουμε το λόγο στον Υπουργό. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Δανό Υπουργό Νίκολας Βάμεν. Αν δεν έχει έρθει, ακόμη θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ιδάλλως πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε με τον Υπουργό. Okay, so he, he should come. Dear colleagues, we have minister here, so we... Έχει καταφτάσει ο Υπουργός. Αν θα θέλατε, λοιπόν να κάτσετε στη θέση σας. Yes.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε διότι ο υπουργό έχει να προλάβει μια πτήση και γι' αυτό δεν μπορούμε να υπερβούμε το χρονοδιαγραμμά μας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 6 το απόγευμα με τη συνεδρίαση. Γι' αυτό και δεν διακόπτω καθόλου τη συνεδρίαση. Καλωσορίζω τον Υπουργό. Όπως ξέρετε παραδοσιακά στα τέλη κάθε προεδρίας ε, υποδεχόμεθα τους υπουργούς και γι' αυτό γίνεται το Μάιο γιατί τον Ιούνιο θα ήταν δύσκολο διότι πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκό συντονισμός ε, δεν είναι μόνο τα θέματα συνοχής, γι' αυτό ήταν δύσκολο να γίνει τον Ιούνιο αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Δίνω το λόγο λοιπόν στον Υπουργό. Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας ευχαριστήσω, εσάς προσωπικά κυρία Πρόεδρε που μου διαθέτετε χρόνο στη σημερινή βεβαρημένη μερισιά διάταξη επιτροπή σας. Θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για τον επικοδομητικό και ανοιχτό διάλογο που είχαμε τους τελευταίους αυτούς μήνες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει έναν σημαντικό και με τα προσθέτω και επικοδομητικό, θετικό ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας νομοθετικής και με πολύ χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την κατάσταση των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο μόλις ένα μήνα πρωτού δώσουμε τη σκητάλη στους ε, Κύπριους φίλους μας. Μετά την ε, εισαγωγή μου, νομίζω ότι έχουμε χρόνο για μια ανταλλαγή απόψεων, στην οποία και προσβλέπω. Αγαπητοί συνάδελφοι, με την αδειά σα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις συνθήκες από τις οποίες έχουμε αναλάβει την προεδρία. Οικονομική κρίση, η οποία ε, πλήττει τις περισσότερες χώρες και αυτό έχει κάνει και τους πολιτικούς και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνούν ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη που θα μπορεί να λάβει μακρόπνοες αποφάσεις και αυτό τάχιστα, με καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Μια τέτοια Ευρώπη πραγματικά νομίζω ότι έχει αναδυθεί μπροστά στα μάτια μας με την ε, οικονομική αυτή κρίση. Τους τελευταίους έξι μήνες, μόλις τους ε, έξι τελευταίους μήνες, 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, που έχει σημαντικές επιπτώσεις ε, και στη δημοσιονομική πολιτική και στη δημοσιονομική πειθαρχία των κρατών μελών. Ένας μόνιμος ε, μηχανισμός σταθερότητας επίσης ε, για τη χορήγηση χρηματοοικονομικής βοήθειας στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης έχει θεσπιστεί έχει συμφωνηθεί ένα μεγάλο επίσης σχέδιο διάσωσης για τη βοήθεια της Ελλάδας και στις 17 του μηνός αποφάσισαν να ενισχύσουν και το τείχος προστασίας ε, οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Βέβαια χρειάζονται και έχουν ήδη ξεκινήσει σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο που θα συμπληρώσουν ε, τα μέτρα που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει ξεκινήσει επίσης διαδικασία για την εκπόνηση ενός συνολικού πακέτου προσανατολισμένου προς την ανάπτυξη με πρωτοβουλίες που θα συμφωνηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Αυτή ήταν η προσέγγιση της Προεδρίας μας για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης. Πρέπει να βαδίσουμε και στα δύο πόδια, δηλαδή να συνδυάσουμε τα απαραίτητα μέτρα δημοσιονομική εξυγίανση και πειθαρχία με διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει και στοχευμένε πρωτοβουλίε για την ε, τόνωση της ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Αυτά τα σημαντικά βήματα έρχονται να προσθεθούν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα κράτη-μέλη της έχουν αναγνωρίσει ότι η απάντηση στις σημερινές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουμε είναι περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη Ίσως μας διδάξει και η ίδια η ιστορία ότι οι εθνικές κυβερνήσεις συνήθως ακολουθούν το μονοπάτι του προστατευτισμού, του εθνικισμού και της ομφαλοσκόπησης ε, όταν ε, υπάρχει ύφεση στην οικονομία. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη φορά αυτό δεν συνέβη. Ξεκάθαρα δεν συνέβη αυτό. Αντιθέτως, η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με πιέσεις από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ενίσχυσε την αλληλεγγύη, την πειθαρχία, αλλά και τη συνεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση δεν έχει δημιουργήσει νέους ε, ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά έχει ενισχύσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε σημαντικού τομείς πολιτικής, διότι αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν η μόνη επαρκής απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Και αν σκάψουμε λίγο πιο βαθιά και διερωτηθούμε γιατί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να ενισχύσουν το ευρωπαϊκό σχέδιο και δεν ε, επιδίωξαν μόνο εθνικούς στόχους, πιστεύω ότι η απάντηση είναι η εξής. Διότι οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τέτοια διασύνδεση μεταξύ τους, είναι τόσο ολοκληρωμένε και διασυνδεδεμένες σήμερα που δεν υπάρχουν άλλε βιώσιμε λύσει, παρά μόνο οι κοινέ δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει απλά άλλη λύση, άλλος δρόμος. Οι οικονομίε μας, οι εταιρείε μας, αλλά και οι λαοί μα εξαρτώνται τόσο πολύ ένα από τον άλλο πλέον, που οι παροχημένες και ε, ομφαλασκοπούσες πολιτικές των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων έχουν γίνει πλέον παροχημένες και απαρχιωμένες. Αντίθετα, όταν δρούμε συντονισμένα, όπως συνέβη για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουμε ε, μία δυνατότητα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των αγορών και να επιτελέσουμε πρόοδο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι μια θετική και ενθαρρυντική εξέλιξη. Και εμείς ως Προεδρία θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στο υπόλοιπο του εξαμήνου για να αυξήσουμε αυτή τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρά ενωμένη και να δίνει αυτά αποτελέσματα που θα βελτιώσουν τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Η Δανική Προεδρία παραμένει προσιλωμένη σε μια ατζέντα, σε ένα θεματολόγιο που θέλει να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Και όπως ε, φαντάζεστε η προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης απαιτεί ε, προσπάθειες ευρύτατες οι οποίες εξαπλώνονται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν τις διαπραγματεύσεις ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Δανική Προεδρία εργάζεται σκληρά για τη δημιουργία συνένεσης υπέρ Τη εκχώρηση ενό μεγαλύτερου μεριδίου του προπολογισμού σε τομεί όπω είναι η έρευνα, η παιδεία, η ενεργειακή απόδοση και οι πράσινες τεχνολογίες. Ταυτόχρονα διαπραγματευόμαστε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης διαφόρων τομεακών πολιτικών με στόχο να πετύχουμε ώστε να το περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση. Δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες εβδομάδες από τη Eurostat. Συνολικά 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι κάτω των 25 είναι άνεργοι. Είναι άνεργοι. Στην Ισπανία και στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας ε, των νέων υπερβαίνει το 5%. Και φυσικά αυτά τα αριθμητικά στοιχεία ε, προκαλούν ε, φόβο και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί πρέπει τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει πιο σταθερές, στεναρές πολιτικές υπέρ της απασχόλησης. Διότι πρέπει να απομακρύνουμε ε, τις ε, πολύ αρνητικές προοπτικές. Ως ηγέτες, ε, ως μέλη της κυβέρνησης, κάνουμε ό,τι μπορούμε και πιστεύω θα αποτρέψουμε αυτά τα τρομακτικά σενάρια. Τι δυναμικό υπάρχει λοιπόν για το μέλλον ε, τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή. Πριν από τέσσερι μήνε είχα την ε, δυνατότητα και την ευκαιρία να συναντηθώ με εσά και να συζητήσουμε μαζί το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή. Όταν έφυγα από την αίθουσα, από τη συνάντηση, ήμουν πεπισμένο ότι από κοινού Συμβούλιο και Κοινοβούλιο μπορούν να θέσουν τα θεμέλια για ε, μια εστιασμένη πολιτική συνοχή που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία θέσεων εργασία, για τη δημιουργία ανάπτυξη από τι δύσκολε αυτέ οικονομικέ συνθήκε. Ταυτόχρονα, έχει ζητηθεί και από του δικαιούχου να είναι πιο απλή στην εφαρμογή τη πολιτική συνοχή αλλά να είναι και παρκώς ελαστική και ευέλικτη για να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η κατάσταση στα κράτη-μέλη, αλλά και εντός των κρατών μελών, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Επίσης, αν τίποτα έχει να μας διδάξει αυτή η κρίση και αν μάθαμε κάτι από αυτή την κρίση, είναι ότι αλλάζουν δραματικά οι συνθήκες, οι καιροί και σήμερα μπορώ να σας αναφέρω και να βεβαιώσω ότι σωστά έτρεφα αυτή την αισιοδοξία και δικαιολογημένα. Είμαι πολύ ε, ικανοποιημένος που καταφέραμε να συμφωνήσουμε των τελευταίων τροπολογιών ε, ε, του κανονισμού και έχουμε συμπεριλάβει στην πολιτική συνοχή μέτρα για τον επιμερισμό των κινδύνων. Θα ήθελα ε, με την ευκαιρία αυτή να αναγνωρίσω και να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για την πολύ βοηθητική και επικοδομητική στάση που τήρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα, γιατί από κοινού καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την νομοθετική διαδικασία έγκαιρα και ελπίζουμε ότι η κρίση που έχει πλήξει τα κράτη-μέλη ε, ε, θα αντιμετωπιστεί με τη σωστή χρήση αυτών των εργαλείων από τα κράτη-μέλη. Η Δανική Προεδρία έχει αναλάβει το καθήκον επίσης της πρόθεσης των διαπραγματεύσεων επί της νομοθετικής θέσμης μέτρων. Με την στήριξη των κρατών μελών, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Απρίλιο κατάφερε μια μερική ε, προσέγγιση ε, σε έξι δαπραγματευτικά ζητήματα που ήταν η εξάντερεσιμότητα, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση και τα μεγάλα σε σχέδια. Επίσης η ευελιξία, η αποδοτικότητα είναι λέξεις κλειδιά που περιγράφουν την προκατρατική συμφωνία για αυτά τα έξι μπλοκ, για τις έξι ομάδες μέτρων. Πριν περάσω στη διαδικασία που θα οδηγήσει ε, στο Γενικό Συμβούλιο των Τελών του Ιωνίου που θα συζητήσουμε το νομοθετικό πακέτο για δεύτερη φορά, θα ήθελα να σας πω λίγα παραπάνω για αυτά τα ε, που μόλις προανέφερα. Αν δείτε το συμβαστική πρόταση και τον προγραμματισμό θα δείτε πώς έχουμε ε, προχωρήσει. Γιατί εκεί αποφασίζουμε πώς ε, εξελίσσονται τα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία επικεντρώνονται γύρω από τους στόχους των δικαιούχων και αποδεκτών. Πρώτον είναι οι στόχοι, δεύτερον τα μέσα. Τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και αυτό χωρίς να πρέπει να επανυποβάλλουν κάθε μία λεπτομεριακή αλλαγή ε, προς έγκριση από την Επιτροπή, μια διαδικασία που είναι σίγουρα χρονοβόρα και θα προκαλέσει καθυστερήσεις στην εφαρμογή. Το ίδιο βλέπουμε και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο. Υπάρχει αποτελεσματικότητα εδώ. Η ε, διαχειριστική αρχή αφενός πρέπει να εξασφαλίσει ότι συγκεκριμένα προγράμματα συνεισφέρουν στην επίτευξη των αναφερομένων στόχων. Αφενός έχει αφετέρου όμω και το καθήκον ε, να αποφύγει τους αχρίαστου ελέγχου που δίνουν στην ε, πολιτική συνοχή, στην φήμη ότι είναι δύσκολο να τη διαχειριστεί κανεί. Έχουμε λοιπόν ε, τεχνικές δαματοληψίας ε, και μέτρα αναλογικότητας. Θα δείτε επίσης ένα συνδυασμό για να έχουμε ευελιξία και αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Συμφωνήσαμε λοιπόν και στο μπλοκ της εξάντε ερεσιμότητας σε σύγκριση με την αρχική πρόταση έχουμε προσαρμόσει τους όρους ε, που είναι πλέον πολύ πιο σωστά στοχευμένοι και άμεσα συνδεδεμένοι στην αποδοτικότητα ε, των δαπανών για τη συνοχή. Δεν είναι μια απλή άσκηση ελέγχου της συμμόρφωσης με τις οδηγίες που τόσο ή άλλως ε, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη διαδικασία παραβάση. Τα ίδια στοιχεία τα βλέπει κανείς και στη συμβαστική πρόταση που έχουμε για τα μεγάλα ε, προγράμματα. Θέλουμε να υπάρχει ένας ανάντια έλεγχος. Θέλουμε να βρούμε εναλλακτικές θετικές προτάσεις ε, και όχι να ε, έχουμε απλά αυτές τις ασκήσεις ελέγχου που γίνονται στα γραφεία από το Συμβούλιο. και επίση θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη να εκμεταλλευτούν και τη μεγάλη εμπειρία τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θέλουμε επίση ε, απλούστευση του κόστου και αυτό το στήριξε το Συμβούλιο. Το ίδιο ισχύει για την ενίσχυση τη παρακολούθηση και τη αξιολόγηση. Και εδώ πάλι βλέπουμε ότι θέλουμε να έχουμε και απλούστευση και αποδοτικότητα. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, με αυτά τα στοιχεία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Απριλίου, έχουμε πλέον ε, θέση στέρεα θεμέλια για μια απλούστευμένη ε, ε, αλλά και πιο αποδοτική μελλοντική πολιτική συνοχής. Και γι' αυτό ζητούμε το Κοινοβούλιο να δεχθεί αυτά τα στοιχεία. Βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Η Προεδρία μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τα μανίκια μας ακόμα σηκωμένα είναι και ακόμη εργαζόμαστε σκληρά μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Και περιμένουμε με ανυπομονησία και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Ιούνιο. Έχουμε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα. Για κάποιες ασκήσεις ε, και επιχείρησεις που ε, θα παράξουν εισόδημα. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε και τις συστάσεις αναχώρα σε σχέση με τον προγραμματισμό. Θα τα δούμε ένα-ένα όλα αυτά. Καταρχά για τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ιδιαίτερα σε ένα τομέα εθνικών, ε, μάλλον σε μια εποχή περικοπών των εθνικών προπολογισμών. Ιδανικά δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να συνεχίσουν την, την πολιτική συνοχή και να, να προσελκύσουν επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, πάντα με απότερο στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης. Βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης τροπολογίας, ε, τροπολογιών της εξαιρετικής πρότασης του Απριλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναγνώριση ευρωπαϊκών προτεραιότητων όπως ε, το Venture Capital για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημειώνουμε καλή πρόοδο και ελπίζουμε να συνεργαστεί και το Κοινοβούλιο και προς αυτό. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις ε, διαδικασίες και τις δραστηριότητε που αποφέρουν έσοδα. Όλοι ξέρουν ότι ο τρέχον κανονισμός είναι δύσκολο στην εφαρμογή του και βάσει μιας καλής πρότασης της Επιτροπής εξετάζουμε δυνατότητα περαιτέρω απλούστευσης, προώθησης ε, της χρήσης ε, των flat rates σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Αυτό θα αποτελέσει όχι μόνο απλοποίηση, αλλά θα αυξήσει και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής. Θα πρέπει εξ αρχής να τεθούν οι σωστοί κανόνες. Αυτό θα δώσει κίνητρα σε μια γενιά εσόδων και θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τους πόρους της συνοχής για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. και θέλουμε να προωθήσουμε και τη συμπράξη διδικού και δημοσίου τομέα γιατί αποτελούν ένα α, τρόπο καλύτερης αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος. Κατά τρίτον, θεματική επικέντρωση, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην πρόταση του νέου κανονισμού. Όλοι συμφωνούν με την ε, ανάγκη να επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα, να μην δισκορπιστούν τα χρήματα αυτά, να χρησιμοποιηθούν για ζητήματα στρατηγικής σημασίας, ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης, δημιουργία θέσεων εργασία. Γίνονται διαπραγματεύσει βάσει τη πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εστιαστούν οι δαπάνε στην κοινοτομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ε, περιορισμό της αλλαγής του κλίματος. Η πρόκληση θα είναι να υπάρχει απαραίτητη ευελιξία όπου χρειάζεται, χωρίς να αποδυναμωθεί ωστόσο ο κανονισμός. Αυτό αποτελεί ε, άγουσα γραμμή. Και από την πλευρά αυτή υπολογίζουμε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Στη γνωμοδότηση του Απριλίου προς το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη στα διαφορετικά τις συμμορφίες ε, των κρατών μελών, ελήφθησαν υπόψη και οι συμφωνίε εμπορική σχέση, Θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και χαίρομαι Συνάδελφοι, να σα αναφέρω ότι οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο χαρακτηρίζονται από την κοινή επιθυμία οι κανόνε την επόμενη προγραμματική ε, περίοδο να καταστούν πιο ε, ισχυροί προ το συμφέρον τη πραγματική οικονομίας. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ και με την Πολωνική Προεδρία και με την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να επαναλάβω το θαυμασμό μου για τη σκληρή δουλειά της Πολωνικής Προεδρίας, γιατί ποτέ δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φανταστεί να έχει προηγηθεί καλύτερη Προεδρία. Θα ήθελα παράλληλα όμως να εκφράσω την αισιοδοξία μου ότι η επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει τις επιτυχίες του προηγούμενου έτους. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την καλή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Προεδρίας μας σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής συνοχής. Ήταν πολύ καλές οι συναντήσεις μας και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την στενή και επιτυχή μας συνεργασία κατά τη διάρκεια της Ιστανική Προεδρίας. Ήταν επικοδομητική η στάση τους για την εξέβρεση βιώσιμων συμβιβασμών. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό Άρα κυρίες και κύριοι, στη θερμή αυτή η μέρα που μοιάζει καλοκαιρινή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και ανυπομονώ να ακούσω σχόλια και ερωτήσεις εκ μέρους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Να ξεκινήσουμε με τον Λαμπέρ, την Κωνσταντσε και μετά αν θα θέλατε, όλοι σας να μου πείτε τώρα ότι θέλετε το λόγο για να μπορέσω να διαιρέσω το διαθέσιμο χρόνο. Ο Λαμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την πολύ ζωηρή σας παρουσίαση και θα πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη που είμαστε κάπως κουρασμένοι. Βλέπετε, ξεκινήσαμε στις 9 σήμερα το πρωί με τον Γενικό Κανονισμό Ψηφοφορίες, Ακρόαση για την έρευνα και την ανάπτυξη και η συνέργεια με τα περιφερειακά ταμεία, άρα πραγματικά μας δώσατε ε, μια νέα ορμή με την ε, ομιλία σας, με την παρουσία σας. Οι σχέσεις ήταν εξαιρετικές, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν ε, άγγιξαν το περιεχόμενο. Ήταν καλές οι σχέσεις μας, αλλά δεν υπήρχαν διαπραγματεύσεις για τα πιο πολλά θέματα στην ε, Επιτροπή μας άλλη άποψη της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, άλλη άποψη του Συμβουλίου. Η συνεργασία θα μπορούσε να είναι καλύτερη, νομίζω. Τουλάχιστον τώρα στις 9 Ιουνίου θα αποκρισταλαθεί η άποψη του Κοινοβουλίου και θα θέλαμε αυτό το θέμα να το συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Σήμερα συναντηθήκαμε και με τον Επίτροπο. Ρωτήσαμε τον Επίτροπο πόσο έχει προχωρήσει, κατά πόσο έχει κάνει συμφωνίες με το Συμβούλιο. Μας είπε ότι όχι, δεν έχουν γίνει συμφωνίες με το Συμβούλιο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει στην πρότασή της, αυτήν η σαφή θέση, και από τις δύο πλευρές και από πλευράς του Κοινοβουλίου και από πλευράς του Συμβουλίου έχει σημειωθεί πραγματική πρόοδος. Πολύ σωστό αυτό και από πλευράς σας και από πλευράς μας, αλλά μπορούμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, επί του συνόλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να ξέρουμε τη θέση μας. Για πρώτη φορά είμαστε σε πλήρη διαδικασία συναπόφασης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Άρα, να πω, ίσως όχι στην Δανική Προεδρία, να πω στην Κυπριακή Προεδρία ότι ας περάσουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε σήμερα το πρωί. Πώς ε, το... οι διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, συνδέονται με τις αρμοδιότητες ε, της Επιτροπής μας. Το γνωρίζουμε το ζήτημα αυτό δεν έχουν καθησυχαστεί οι ανησυχίε του Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου, γιατί κανεί δεν ξέρει τι θα γίνει στα τελικά συμπεράσματα τον Ιούνιο. Το negotiation box είναι black box. Είναι μαύρο κουτί. Δεν ξέρουμε τι του έχουν βάλει μέσα για θέματα αρμοδιότητας του κανονισμού μας. Μπορεί τελική ανάλυση να έχουμε λίγο προβλήματα στα θέματα των αρμοδιοτήτων. Μήπω μπορείτε να σχολιάσετε. Δίκιο έχει ο κύριος Χάν. Είναι ανοιχτή η διαπραγματεύση η οποία επίκειται όλη τη ύλη. Για πείτε μας. Και κατά τα άλλα συμφωνώ απόλυτα για το σημαντικό έργο και τον επαναπροσανατολισμό σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά προβλήματα για τις επερχόμενες επενδύσεις στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης που πρέπει να συμβούν. Είναι σημαντικό τον Ιούνιο η πολιτική συνοχής με όλα τα εργαλεία της να είναι βιώσιμη και εφαρμόσιμη, γιατί είμαστε όχι μοναδικός, αλλά ένας πολύ σημαντικός φορέας επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη, που μπορούν να μας προχωρήσουν μπροστά. Και αυτά είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα χέρια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ερωτότητα. Και γιατί σε πολλές περιπτώσεις ακούμε και στο ιστορικό αλλά και στο εξωτερικό του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα κονδύλια. Μα τα κονδύλια είναι σημαντικά. Υπάρχουν χώρες των οποίων οι επενδύσει το μεγαλύτερο τμήμα τουλάχιστον, προέρχονται από τα διευθυντικά ταμεία στην παρούσα φάση. Άρα, σε ό,τι αφορά ένα περιεκτικό κείμενο, τον... μάλλον σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, θα θέλαμε ένα θερμό κείμενο από το Συμβούλιο τον Ιούνιο. Η Κωνσταντζα Κρέλε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πολύ πιστική η παρουσίασή σας και χαίρομαι ιδιαίτερα Μιλήσατε για τις δύο πλευρές, ε, τις δύο διαφορετικές πολιτικές, πλευρές της πολιτικής συνοχής. Αυτό που διαπραγματευόμαστε στο Κοινοβούλιο, το νομοθετικό πακέτο, αλλά και την χρηματοδοτική διάσταση, γιατί χωρίς χρήματα μπορεί να θέλουμε ότι θέλουμε εμείς στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Από την παρουσίασή σας συμπεραίνω ότι υπάρχει μια αλλαγή ε, ίσως ε, νοτροπία στο Συμβούλιο, υπό την έννοια ότι αναγνωρίζουμε ότι τα χρέη και η οικονομία, η εξοικονόμηση χρεών είναι φυσικά ένα σκέλος, αλλά ένα άλλο σκέλος είναι ε, η παροχή κινήτρων ανάπτυξης. Και αν προχωρήσω και ένα βήμα παραπέρα, το μοναδικό το, με το οποίο μπορούμε να δώσουμε τέτοια κίνητρα ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πολιτική συνοχής. Άρα θεωρώ μετά από τα λόγια που άκουσα ότι θα δεσμευτείτε, θα ταχθείτε στο υπόλοιπο της Προεδρίας σας, αλλά και τον καιρό που θα είστε ένα απλό μέλος του Συμβουλίου, προκειμένου η πολιτική συνοχή να λάβει το κατάλληλο προϋπολογισμό τον οποίο πρότεινε το Κοινοβούλιο. Γιατί πρόκειται για μια σκόπιμη και φύ, ε, αν θέλετε, μέθοδο ε, δαπάνης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το δεύτερο σημείο τώρα, το τι μπορούμε να... και τι πρέπει να διαπραγματούμε στο μέλλον από κοινού το περιεχόμενο διαφορετικών κανονισμών, γιατί πέρα από το γεγονός ότι τα black boxes παραμένουν black boxes, μαύρα κουτιά, ε, ακούμε, ακούμε ότι γίνονται και υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις και μπορώ να φανταστώ ότι με κάποιες από τις προτάσεις του Συμβουλίου κάπως γρήγορα θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να αναπτύξουμε κάποιες κοινέ αντιλήψεις. Θεωρώ λοιπόν ότι για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε αλλά και σε θέματα performance reserve και σε πολλά άλλα θέματα. Ως εκ τούτου, είναι σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και ασφαλώς υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία δεν ε, συγκλίνουν οι απόψεις μας. Ξεκινάμε από τον κώδικα της διοντολογίας σε ό,τι αφορά τις ε, συμβάσεις εταιρικών σχέσεων και στην αποδυνάμωση τους ε, σε agreements, σε συμφωνίες, σε ό,τι αφορά την εξάντερησιμότητα Πρέπει να πω ότι οι δηλώσεις του Συμβουλίου είναι κάπως ε, διφορούμενες. Από τη μία είναι υπέρ, από την άλλη διαγράφονται και ολόκληρα τμήματα σε ό,τι αφορά την οριζόντια εξάντε αιρεσιμότητα σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, της ε, απαγόρευσης των διακρίσεων, τα άτομα με αναπηρία, όλα αυτά θέλετε να διαγράψετε, όλα αυτά μας δυσκολεύουν, καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα καταφέρουμε μέσω της ε, διαπραγματευτικής οδού να βρούμε κοινό τόπο προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα κοινό στόχο. Αν είναι δυνατόν αυτά τα διαπραγματευτικά μαύρα κούτια να καταφέρουμε να τα διαπραγματευτούμε στα πλαίσια της συναπόφασης. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση να μην προκύψει ένα μεγάλο μαύρο κουτί το οποίο θα είναι αδιαπραγμάτευτο από πλευράς του Συμβουλίου. Αυτό δεν θα είναι φυσικά αποδεκτό γιατί δεν θα συνάδει και με τις συνθήκες και το ξέρω ότι δεσμευτήκατε ότι θα τηρηθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και θα ήθελα παρακαλώ να τηρήσετε το λόγο σας γιατί νομίζω ότι είναι Προ το συμφέρον μα να αναπτύξουμε μια σύγχρονη πολιτική συνοχή, η οποία στην τελική ανάλυση θα ωφελήσει όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Και νομίζω ότι αυτό που θέλει να πετύχει και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα μας ε, οθήσει σε μια καλή συνεργασία για το μέλλον. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, επόμενο να είναι συντομότερο προηγούμενο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Μάνερ έχει πάρει το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ τον Υπουργό για την εξαιρετική του τοποθέτηση. Όπως είπαν και οι προλήσατες, είναι πολύ σημαντικό να ακούει κανείς ότι η πολιτική συνοχή είναι πολιτική επενδύσεων ε, εν τέλει. Και ελπίζω να κρατήσετε αυτή τη γραμμή και στο Συμβούλιο και να υπερασπιστείτε την πολιτική ε, συνοχή ε, και στι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό. Συμφωνώ με τον κύριο Βενιστερόη. Έχουμε λάβει πολλέ πληροφορίε για όσα λαμβάνουν χώρα στο Συμβούλιο, όμω κάποιε λεπτομέρειε θα μπορούσαν να γίνονται καλύτερα κάποια πράγματα ε, επιμέρους θα έλεγα πρέπει να διαθετηθούν αναφέρουμε στις επιμέρους σχέσεις ε, του Συμβουλίου με κάποιους εισηγητές μας. Σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θέλω να καταλάβω ποιο είναι το γενικότερο αίσθημα στο Συμβούλιο ε, σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα. Κάποια κρατηβέλη επιθυμούν μία οριζόντια περικοπή του ευρωπαϊκού προλογισμού κατά 10%. Εσείς ακριβώς πώς θα υπερασπιστείτε την πολιτική συνοχή μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες προβληματικές, αν θέλετε, ζώνες στην στο Συμβούλιο και θέλω να ακούσουμε κάποια στοιχεία ε, από εσά η Πρόεδρος. Καλύτερα να απαντήσετε σε αυτά τα τρία ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, και μετά να συνεχίσουμε. Βεβαίω, κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα σα ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια, για την εισαγωγική μου τοποθέτηση. Πραγματικά ε, το εκτιμώ ιδιαίτερα. Κύριε Βανιστερόη, είπατε ότι μπορούμε να τηλήσουμε διδάγματα από αυτή την εμπειρία ώστε να έχουμε καλύτερη συνεργασία στο μέλλον. Αυτό είναι μάλλον αλήθεια. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές ε, ειλικρινώς πώς κινούμεθα, αλλά όλοι μπορούμε να αντιλήσουμε διδάγματα και ε, η Δανική Προεδρία μπορεί να αντιλήσει διδάγματα και να περάσει κάποια μηνύματα στην απερχόμενη Προεδρία του Συμβουλίου. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει και ένας κύκλος στη διαδικασία λύσης αποφάσεων, η διαπραγματεύση για το πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο. Το δημοσιονομικό κουτί όπως έθιξαν και κάποιοι από τους αγορητές, είναι ένα μαύρο κουτί. Εγώ διαφωνώ αν θέλετε με αυτό το νόρμα, αυτή την περιγραφή, όμως... Επειδή δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή και έχουμε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο για αυτό το ζήτημα, θέλω να ενημερώσω την Επιτροπή σας ότι πριν από κάθε συνεδρία του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων έχουμε συνάντηση με εκπροσώπους του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την εποπτεία του κυρίου Λαμασούρ. Ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο σε ποιο σημείο έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσει και μεταφέρουμε έπειτα το μήνυμα του Κοινοβουλίου στο ίδιο τραπέζι των συζητήσεων. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια διάδραση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Προεδρία και το Συμβούλιο. Και αισθάνομαι ότι μπορώ ειλικρινά να πω ότι δεν έχει υπάρξει προηγούμενη Προεδρία που να έχει πιο στενή συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων και αισθάνομαι περήφανος γι' αυτό. Και σημάδι αυτή τη στενή συνεργασία που θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε καθώς θέλουμε να είναι έτοιμο το διαπραγματευτικό κουτί, ώστε να το συζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής στα τέλη Ιουνίου. Ταυτόχρονα συνειδητοποιούμε και απαντώ και στην κυρία Κρέιλ ότι για μας ε, είναι σαφές. Η διαδικασία της συναπόφασης ισχύει προκειμένου και σίγουρα θα πρέπει να σεβαστούμε τους θεσμούς, τα θεσμικά όργανα, τους συνομοθέτες Άρα και το Συμβούλιο, και το Κοινοβούλιο, αλλά βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως το Κοινοβούλιο κάποια στιγμή θα έρθει και θα αρθρώσει λόγο και θα μας παρουσιάσει την διαπραγματευτική του θέση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αντίστοιχα θα πρέπει να διαρθρώσει τη θέση του Συμβούλιο. Και μιλώ για διαπραγμάτευση και δεν το κάνω τυχαία, διότι αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι συμπεφωνηθέντας το Συμβούλιο δεν είναι η τελεία και παύλα αν θέλετε στο θέμα. Μετά την θέση του Συμβουλίου έρχονται οι με το Κοινοβούλιο. Αυτό προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να σεβαστούμε ο ένας το ρόλο του άλλου. Αυτό είναι σαφές. Ταυτόχρονα θα πρέπει και το ίδιο το Συμβούλιο να καταλήξει πρώτα απ' όλα στη διαπραγματευτική του θέση πριν ε, ξεκινήσει τη με το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή σειρά των πραγμάτων. Και να περάσω στο επόμενο σημείο, σχόλιο που ακούστηκε. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο κατά διαθερωτικά, τα μια συνοχή, συγγνώμη, για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Μα ναι, βεβαίως. Πολλά από αυτά τα project όμως ήδη έχουν παράξει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Και επίσης είμαι της γνώμης ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μας και να ρωτηθούμε μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από ό,τι κάναμε στο παρελθόν. Και εγώ περιμένω από τη δική επιτροπή και από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν να πούνε ναι, μπορούμε να είμαστε καλύτεροι ώστε να δαπανούμε το κάθε ευρώ με καλύτερο τρόπο, στα κατάλληλα project, ώστε η απασχόληση και η ανάπτυξη να χρησιμοποιηθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι η κοινή μας ευθύνη. Γι' αυτό η Δανική Προεδρία είναι πάρα πολύ ευτυχής, γιατί ακολουθείται αυτή η παράλληλη διτή διαδικασία. Δεν μιλούμε μόνο για λιτότητα. Δεν είναι μόνο να σφίγγει στο ζωνάρι σημαντικό, αλλά πρέπει να δημιουργήσει τις εργασίες και ανάπτυξη. Δεν μπορεί το ένα να λειτουργήσει χωρί το άλλο. Υπ' αυτή την έννοια. Το να σηκώσει αν θέλετε τα μανίκια η Ευρώπη Getting Europe at Work ήταν το σλόγγαν της Δανικής Προεδρίας. Είναι κάτι που πραγματικά εκφράζει σε μία φράση το πνεύμα μας. Κύριε Μάνερ, είπατε ότι υπάρχουν διαφωνίες στο Συμβούλιο. με τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Αν κατάλαβα καλύτερα την ερώτησή σα. Και που υπάρχουν διαφωνίε για τι περικοπέ και τι μπορούμε να περιμένουμε για την πολιτική συνοχή. Κοιτάξτε, η Ιδανική Προεδρία ήταν έτοιμη να βάλει και αριθμητικά στοιχεία στο διαπραγματευτικό κουτί. Αλλά αυτό που ακούσαμε από την πλειοψηφία των κρατών μελών και από την Κομισιόν, αλλά και από του εκπροσώπου του Κοινοβουλίου, ήταν ότι είναι πρόωρο αυτή τη χρονική στιγμή να βάλουμε και αριθμητικά στοιχεία στο διαπραγματευτικό κουτί. Οπότε το δεχτήκαμε και γι' αυτό δεν θα υπάρξουν. Θα δοθεί λοιπόν πιο πολύς χρόνος και στο Κοινοβούλιο να αποφασίσει πού θέλετε και πώς θέλετε να επιμερίσει τα κορδίλια και με ε, ποια ποσοστά. Το γεγονό ότι δεν βάζουμε συγκεκριμένα ποσοστά και αριθμητικά στοιχεία στο διαπραγματευτικό κουτί είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μου επιτρέπετε σήμερα να σας πω σήμερα εδώ τέτοια αριθμητικά στοιχεία. Θα υπάρξει ε, μια σχετική έκθεση από την Κυπριακή Προεδρία εν ευθέτω χρόνο. Εμείς θα καταλήξουμε σε ένα συνολικό, εμπεριστατωμένο, διπραγματευτικό κουπτί χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί θα έρθουν από την Κυπριακή Προεδρία. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω κάτι για περικοπές σε σχέση με την πρώτα, περαιτέρω περικοπές σε σχέση με την προτείνη Κομισιόν και σε τι βαθμό. Πάντως δεν είναι μυστικό ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν δύο βασικές θέσεις. Οι μεν θεωρούν ότι είναι καλή πρόταση Κομισιόν και δεν θα μπορούσε να συμφωνηθεί ούτε ένα ευρώ λιγότερο. Και από την άλλη, κάποιοι που θεωρούν ότι είναι υπερβολικά υψηλή πρόταση κατά 100 δις. Και σήμερα το πρωί που συζητούσαμε το ίδιο θέμα, οι θέσει είναι σαφεί, σταθερέ και ο κανένας δεν μετακινείται. Θα υπάρξει λοιπόν μάχη μέχρι το τέλος. Μάχη μέσα στους κόλπους του Συμβουλίου και μετά μάχη ανάμεσα στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Δεν εκπλήσει κανένα αυτό. Δεν θα γίνει όμως η μάχη κατά τη Δανική Προεδρία, αλλά κατά την Κυπριακή Προεδρία. Διότι το δικό μας καθήκον, αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς, είναι, να, ε, είναι έτοιμο το διαπραγματευτικό κουτί τον Ιούνιο, ώστε να επιτρέψουμε στους Κυπρίους συναδέλφους μας να ολοκληρώσουν αυτή τη δουλειά στο δεύτερο ημίση τη χρονιάς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος. Πέντε ακόμη αγορητές έχω στο καταλογό μου. Αν θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τις απαντήσεις του Υπουργού, μόνο ένα λεπτό αναομιλητή. Κύριε Λεφόνση, θέλετε το λόγο. Τρεις ομιλητές τελικά, κάποιοι υποχωρούν, ενάμιση λεπτό. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Φλάσακ, εκτιμώ τις προσπάθειές σας ε, να πλουστεύσετε την πολιτική συνοχή και να βελτιώσετε την ευελιξία, ιδίως ό,τι αφορά τη διανομή των κονδυλίων μεταξύ των ε, αναπτυγμένων, μη αναπτυγμένων και πολύ αναπτυγμένων περιοχών. Μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη ελαστικότητα πάνω και από το 10%. Δεύτερη ερώτηση. Η μέθοδος Leader φάνηκε να είναι αποτελεσματική στα περιοργία ζητήματα. Θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς Μια μελλοντική κατεύθυνση λοιπόν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη συμμόρφωση με τις στρατηγικές που χαράσουν ίσως οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ιάννα Μιράντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, οι εξηγήσεις που μας δώσατε για την συμμετοχή των περιφερειών η δομή που είναι διαφορετική στα κράτη-μέλη. Ε, δεν με πείσατε ιδιαίτερα γιατί δεν μας δώσατε συγκεκριμένα στοιχεία. Να ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος. Ε, έχουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης όμως. Ποιες είναι οι διαφορές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο στο πλαίσιο της εκπροσώπησης ε, των ε, διαφορετικών εδαφικών επιπέδων στα κράτη-μέλη. Θεωρείται ότι πρέπει να συμμετέχουν οι περιφέρειες σε όλα τα στάδια ε, της, μέχρι δηλαδή την παρουσία και την αξιολόγηση των σχεδίων ή να παραμένουν παρατηρητές, όπως είναι η τάση σε κάποια κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η Μαρία Ριγκόγεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την πλήρη ενημέρωση. Έχω ένα αίτημα και μια παράκληση πιο πολύ ε, στην ε, διάσκεψη κορυφής του Ιωνίου. Έχουμε ελπίδες, ε, πολλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποθέσει ελπίδες τους στο ότι η ευρωπαϊκή πολιτική πλέον θα ξαναβγεί στο προσκήνιο. Συμφωνώ μαζί σας ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση είναι θεμελιώδης σημασίας. Η παράκληση λοιπόν και το αίτημά μου προς τη Δανική Προεδρία θα ήταν να δρομολογήσετε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, ένα ονοδικό χάρτη για τη δημιουργία απασχόλησης ώστε η κρίση αυτή, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε, να γίνει μια ευκαιρία και να μην ε, απογοητεύσει η Δανική Προεδρία τόσους Ευρωπαίους πολίτες που ε, περιμένουν η επόμενη διάσκεψη κορυφή να κλείσει ακριβώς με μια τέτοια πρόταση, με έναν οδικό χάρτη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πρόεδρος, αν δεν θέλει κάποιο άλλο το λόγο θα δώσω το λόγο στον Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ. για τα θέματα της ε, κατανόμης επιμερισμού μεταξύ περιφερειών. Έχουμε τις ε, περιοχές ή ε, περιφέρειες μετάβασης και το θέμα είναι καθαρά ποιος πληρώνει για ποιον. Και φυσικά δεν θα σας εκπλήξω ότι διαφέρουν και οι απόψεις. Μάλλον θα συμπεριληφθεί στην τελική συμφωνία αυτό το θέμα, στην τελική συμφωνία για, τη, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αφού σταθμίσουμε τα υπέρ και τα κατά με τα διαθέσιμα μέσα Σήμερα δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο πάνω στο θέμα αυτό, γιατί είναι ιδιαίτερα λεπτό το ζήτημα και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να λάβουμε τι σωστέ αποφάσεις. Αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ όμως είναι ότι με πνεύμα συνεργασίας θα λάβω υπόψη μου τις απόψεις που μου διατυπώσατε σήμερα. Εταιρική σχέση, περιφέρειες. Θέλουμε να έχουμε διαβούλευση με όλους όσους θα φυγούν από τα διάφορα προγράμματα που θα ολοκληρωθούν. Και φυσικά αυτό θα το κάνουμε. Προέρχομαι από μια χώρα ε, που έχει παράδοση στη διαβούλευση, άρα αυτό είναι προφανές. Και υπήρξα μάλιστα δήμαρχος. Έχω διατελέσει δήμαρχος κατά το παρελθόν και γνωρίζω πολύ καλά πόσα μπορεί να κερδίσει το εθνικό επίπεδο να συνομιλεί με το τοπικό και το περιφερειακό. Άρα θεωρώ ότι όσο περισσότερη ενέργεια, μυαλό, καλή διάθεση μπορεί να δημιουργηθεί, θα είναι καλό, διότι θα ήταν πραγματικά μια απώλεια αν δεν ε, περιλάβουμε το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γιατί αυτά τα επίπεδα ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία είναι πολύ κοντά στους πολίτες, γιατί εκεί γίνεται η εφαρμογή. Φυσικά λοιπόν και θα πρέπει να έχουμε αυτές τις διαβουλεύσεις. Ταυτόχρονα τώρα οι εμπλεκόμενοι φορεί, τα κράτη-μέλη όμως επίσης ε, έχουν ε, ένα θεμητό ενδιαφέρον ε, να ολοκληρωθεί αυτή η δυσκίνητη διαδικασία κατά τον πιο ομαλό τρόπο. Επίσης τον Απρίλιο είπαμε ότι θα πρέπει κανονισμοί να λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά εθνικά συστήματα και παραδόσεις να λαμβάνονται υπόψη εθνικές ιδιαιτερότητες δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ισορροπία, τη χρυσή τομή και σίγουρα είναι προς ε, το συμφέρον όλων μας να καταλήξουμε. Το τελευταίο θέμα ε, και ερώτημα, αν η Δανική Προεδρία, η κυρία Ριγκόγεν Πέριθ, έθεσε αυτό το ερώτημα. Αν η Δανική Προεδρία θα καταθέσει στο τραπέζι μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση, δεν θα το κάνουμε μόνοι μας, αλλά θα εργαστούμε πάρα πολύ στενά και με τον πρόεδρο Φον Ρομπέι τι επόμενες εβδομάδες ο δικός μας στόχος, ο δικό μας καθήκον, όπως το έχουν διατυπώσει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, της προάλλης των επίσημη του συνάντηση, είναι σαφές ότι δηλαδή πρέπει να προτείνουμε αυτό το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μία δέσμη μέτρων για την εξασφάλιση τη ανάπτυξη και τη απασχόληση. Και αυτό θα το πράξουμε σε στενή συνεργασία, παραλαμβάνω, με τον πρόεδρο Φων Ρομπέι, διότι πρέπει να δημιουργήσουμε θέσει εργασία. Και ανάπτυξη. Έχουμε 25 εκατομμύρια νέους, των οποίων 5,5 είναι, εκατομμύρια είναι νέοι, όπως προείπα. Ουσιαστικά λοιπόν εδώ κάνουμε αν θέλετε μία δοκιμή, ένα τεστ και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας ανακόψει από τη σωστή δράση. Δηλαδή να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητα με, για προσαρμογή μάλλον, με τη δημιουργία ανάπτυξη και απασχόλησης. Και αυτό θα πράξουμε τι επόμενες εβδομάδες που έχουμε εμεί ακόμη την ευθύνη, αλλά και μετά θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ε, στην τριάδα των ε, χωρών τη Προεδρίας αυτές τις προσπάθειε. Μετά τον Ιούνιο, ελπίζω αν συναντηθούμε να μου πείτε ότι μας ακούσατε και με την συνένωση των δυνάμεών μας καταφέραμε κάτι καλό. Αυτός είναι ο στόχος της Δανικής Προεδρίας και αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Και θέλω να είμαι ξεκάθαρο πάνω σε αυτό. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μα. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων των κρατών μελών, την υποστήριξη τη Κομισιόν, αλλά πάνω απ' όλα την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, να χειροκροτήσουμε και να ευχαριστήσουμε την Προεδρία για την παρουσία εδώ του κύριου Υπουργού. Θέλω να σας πενθυμίσω όμως ακόμη κάτι. Όταν είχαμε συναντηθεί μαζί και με τους συζητητές είχαμε πει ότι πριν το τέλος της ε, ε, Προεδρίας θα έρθει κάποιος να μας ενημερώσει για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες άλλες κοινέ θέσεις, ε, τι έχετε τέλος πάντων επιτύχει ε, συνολικά στην Προεδρία του Συμβουλίου. Ναι, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω θα έρθει ε, ο, Στέφαν ε, που πρέπει να σας πω ότι σήμερα ήθελε να είναι στη θέση μου, αλλά την άλλη φορά θα είναι ο Στέφαν. Εδώ ολοκληρώνει τη σημερινή συνεδρίαση. Αύριο το πρωί σε 9 παρακαλώ να είστε εδώ για τη συνέχεια των εργασιών μας.